Λοιπόν, ε, καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έναρξη. Κάποιος ξέχασε να πει στην Πρόεδρο ότι άλλαξε η αίθουσα της συνεδρίασης και ούτως ή άλλως μας παίρνει πάντα λίγο χρόνο. Για άλλη μια φορά έχουμε μια διαφορετική συνεδρίαση από αυτές που είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες και θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Κανείς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει από πλευρά τη Προέδρου. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε απευθεία στη δημόσια κρόαση σχετικά με την τραπεζική εποπτεία και την εξυγίανση και να δούμε τα επόμενα βήματα. Εγώ δεν θα σας καθυστερήσω άλλο γιατί ούτως ή άλλως ε, μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε το χρόνο που χάσαμε για να κάνουμε πιο χρήσιμη συζήτηση και θα ήθελα να δώσω στους συζητητέ, ε, Κυρίω τη Μαριάν Τάισεν, η οποία κάνει την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Σφεν Κίγκολ, ο οποίο κάνει ε, την έκθεση για το EBA. Μάριαν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ στην αίθουσα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις που έχουμε αναχείρας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο σημαντικά πράγματα. Οι περισσότεροι από τους παρισταμένους είναι ικανοποιημένη διότι επιτέλους έχουμε κάποιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να έχουμε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό εποπτείας που επιτρέπει να έχουμε μέσα για να ε, εξετάσουμε τι καθήκοντα αναλογούν στον καθένα βάσει του συστήματο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Σα υπενθυμίζω την έκθεση Χωσέ Γκαρθία Μαργκάλιο που έγινε πριν από κάποιο διάστημα. Αυτό ο μηχανισμό υποπτία είναι πολύ σημαντικό διότι είναι πολύ σημαντικό να επανακαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Πρέπει να υπάρξει και εκ νέου εμπιστοσύνη στον τομέα και μια μορφή υποπτία τέτοιου τύπου θα μας ε, βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Θα έχουμε λοιπόν ένα μηχανισμό εποπτείας ε, ο οποίος θα μπορεί να ε, εποπτεύει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εξάλλου, από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γνωρίζουμε ότι η δημιουργία αυτού του μηχανισμού αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκια ώστε αυτός ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός, τον οποίο βαφτίσαμε πριν από δύο μέρες, να μπορέσει να ε, εισρεύσει κεφάλαια στις τράπεζες χωρίς να χρειαστεί να περάσει ε, μέσω της Ατλάντα που εδρεύει ο μηχανισμός. Και αυτό φυσικά είναι μια σημαντική αλλαγή. Κάτι ακόμα το οποίο ε, παρατήρησα στις προτάσεις είναι ότι υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία μας ανησυχούν, ε, μας ανησυχούν και με τα οποία συμφωνούν αρκετοί συνάδελφοι. Για παράδειγμα, η πρόταση γίνεται ε, με βασικό ε, μέσο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και υπάρχουν και άλλα 10 κράτη-μέλη φυσικά. Και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των 27, ε, θα πρέπει να δούμε ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλύπτονται. Ε, οι εθνικές τράπεζες, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι το επίκεντρο όλες της διαδικασίας. Τι αρμοδιότητες θα έχουν οι εθνικές τράπεζες και επίσης τι σχέση υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ε, τα, θέμα, τα καθήκοντα εποπτείας που τις αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία του όλου αυτού του μηχανισμού. Πρόκειται λοιπόν για ανησυχίες οι οποίες ανακύπτουν όταν κάποιος διαβάζει αυτό το μηχανισμό. Θα σκεφτεί βέβαια κανείς ότι όλες αυτές οι ανησυχίες απορρέουν από την επιλογή και της νομικής μας βάσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας εποπτείας. Στην πραγματικότητα όμως ο πραγματικός λόγος της ανησυχίας δεν είναι ε, αυτός. Εγώ θεωρώ ότι οι κανονισμοί που έχουμε εδώ και εξετάζουμε και ακόμα και αυτή η διαδικασία που αναθέτει αυτά τα νέα καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούν να προκύψουν ω απάντηση σε όλε αυτέ τι ανησυχίε. Και θα ήθελα να ζητήσω από του εμπειρογνώμονέ μα να απαντήσουν ακριβώ σε αυτό. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Θα ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν όσα έχουν να μα πούν οι εμπειρογνώμονε, γιατί γνωρίζουν τα θέματα πολύ καλύτερα από εμά. Γι' αυτό άλλωστε του αποκαλούμε και εμπειρογνώμονε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω συγκεκριμένε απαντήσει στα θέματα αυτά μέχρι ποιου βαθμού μπορούμε να ε, προχωρήσουμε με αυτό το μηχανισμό εποπτείας. Και αυτό το ως εποπτικός φορέας που θα δημιουργηθεί στη Φραγκφούρτη τι ακριβώς θα κάνει. Ε, θα μπορέσει να καλύψει και τα κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν προκειμένου να έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης. με τη συγκεκριμένη νομική βάση μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα μηχανισμό εποπτείας των 27, ο οποίος ε, ε, θα περιλαμβάνει και μια ρήτρα opt-out, αντί να ξεκινήσουμε με τους 17 με δυνατότητα opt-in για τους υπόλοιπους 10. Ίσως θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια στενότερη συνεργασία μόνο με τα κράτη της Ευρωζώνης. Τώρα, ο κανονισμός για την εσωτερική αγορά για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται παντού οι ίδιοι κανόνες εποπτείας. Πώ θα πρέπει να γίνει το επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Φορέων και των Εθνικών Εποπτικών Φορέων. Έγινε μια κρόαση στις 3 Σεπτεμβρίου και ακούστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, πίνακας. Δεν ξέρω αν κάποιο το επεξεργάζεται, αν το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε εσείς. Και τέταρτον, τι ακριβώς ε, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την άποψή σας. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε επίσης τη διάκριση μεταξύ του νομισματικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εάν η, η πρόταση αυτή περάσει και εφαρμοστεί, ε, τα, καθήκοντα, τα εποπτικά καθήκοντα. Και εδώ ο πρόεδρος Δράγκη μας είπε ότι οι νομικές υπηρεσίες και ε, όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται από αυτού και της Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κι εσείς ε, περισσότερο. Όσον αφορά τώρα τη λογοδοσία θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και να προχωρήσουμε την περαιτέρω. Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα κατά την άποψή μα και θα ήθελα να ξέρω πώ μπορούμε να αυξήσουμε τη λογοδοσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω τι απαντήσει των εμπειρογνωμόνων τώρα. Thank you very much. Uh, and now θα ήθελα να μην επαναλάβω τα ίδια για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που πραγματικά ανταποκριθήκατε τόσο γρήγορα με τέτοια ταχύτητα στην πρόκλησή μας. Είναι πολύ σημαντικό ε, που σήμερα η αίθουσα είναι γεμάτη. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη ε, ένταση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι το γεγονός ε, της δημιουργίας αυτής της Τραπεζικής Ένωσης αντιμετωπίζεται από όλους μας σαν πραγματικά ένας ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας να βγούμε από την κρίση. Το να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε το ρίσκο είναι επίσης ένα καθοριστικό βήμα και σαφώς δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο. Όλοι είδαμε πόσο ακριβό είναι ένα σύστημα εποπτείας των τραπεζών το οποίο δεν λειτουργεί. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να αφήσουμε αυτό το σύστημα με τέτοιες απρόβλεπτες και αρνητικές συνέπειες. Ένα σύστημα εποπτείας των τραπεζών που δεν λειτουργεί είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Το θέμα της κυριαρχίας που πρέπει να την μοιραστούμε με άλλους, το θέμα αυτό βεβαίως μας οδηγεί σε δυσκολίες και προβλήματα. Γι' αυτό και πρέπει να εργαστούμε για όλα αυτά τα θέματα με τρόπο πολύ ουσιαστικό. Πιστεύω ότι όλοι που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι διατεθειμένοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Ποια είναι τα κεντρικά ερωτήματα για μένα. Πρώτον, ποιος θα πρέπει να είναι αντικείμενο αυτής της ενιαίας εποπτείας. Το θέμα των σχέσεων που υπάρχουν επίσης μεταξύ αυτού του επιμερισμού της δύναμης, της πολιτικής ευθύνης και φυσικά της ανάληψης των ευθυνών με την έννοια χρηματοδότηση αυτών των ε, αρνητικών συνεπειών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα με δύο διαφορετικές φάσεις και θα πρέπει να δούμε πώς από τη μία έχουμε την πολιτική δύναμη, την πολιτική ισχύ και από την άλλη την οικονομική ανάληψη ευθυνών. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, πώς οι εμπειρογνώμενες βλέπουν τα νομικά εμπόδια, τα νομικά σύνορα ενδεχομένως για μία εποπτεία η οποία θα ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τον δημοκρατικό έλεγχο. Σήμερα υπάρχει το θέμα της μη ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής. Ο έλεγχος λοιπόν, η εποπτεία, θα πρέπει εδώ να μην προσκρούσει σε νομικά εμπόδια. Δεύτερο ερώτημα που επίσης αποτελεί περιορισμό. Εάν βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια νομικά εμπόδια και σύνορα, οι χώρες οι οποίες τελικά θα συμπεριληφθούν στο σύστημα αυτό θα πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες σχέσεις με τις χώρες εντός και εκτός του ευρώ. Εδώ βλέπουμε ότι ο κανονισμός, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέτει πολύ συγκεκριμένους ε, όρους όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν ιδιαίτερα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης και των κρατών που είναι εκτός Ευρωζώνης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτή αυτός ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας θα αντιμετωπίσει το θέμα της κυριαρχίας και αυτού του ελέγχου και της ε, διαφορά τη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει σήμερα στην διαδικασία λήψη αποφάσεων μεταξύ των χωρών του ευρώ και των άλλων χωρών. Οι εμπειρογνώμονε πώ αντιμετωπίζουν την πρόταση τη Επιτροπή όσον αφορά την ίση μεταχείριση των χωρών που θα βρίσκονται εντό και εκτό αυτού του μηχανισμού. Επίση, πώ βλέπουν ε, την, ε, το θέμα των δικαιωμάτων λήψη αποφάσεων. Πώς, ε, αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό όσον αφορά το σημερινό ισχύον σύστημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει περιθώριο ελιγμού, ναι ή όχι. Και τι επιπτώσεις βλέπετε, αν πραγματικά ε, περάσουμε σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Τέλος, όσον αφορά την ΕΙΜΠΑ, και τον κανονισμό. Πώς βλέπετε τους κανονισμούς, πώς αντιμετωπίζετε εσείς τους κανονισμούς ε, για την λήψη αποφάσεων και την ψηφοφορία. Είναι ικανοποιητικό το σύστημα που προσφέρεται από τη στιγμή που ο ενιαίος μηχανισμός υποπτίας φυσικά ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας, στην ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των κρατών που θα ενσωματωθούν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και των άλλων. Βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη να συμπληρωθεί ο παρόν κανονισμός με επιπλέον μέτρα και υποχρεώσεις. Γιατί πριν περάσουμε στα περαιτέρω στρες τεστ των τραπεζών, μήπως θα έπρεπε εκ των προτέρων να θέσουμε κάποιους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και συμπεράσματα από την παρούσα εμπειρία, από την μέχρι τώρα εμπειρία μας από την κρίση. Θα ήθελα να μου πείτε πολύ συγκεκριμένα τι θα πρέπει κατά την άποψή σας να αλλάξει στον κανονισμό ΕΒΑ. Uh, we need to try and stick within our, our minutes time. Ευχαριστώ. Να τηρήσουμε το πεντάλεπτο, για να μην χάσουν χρόνο στο τέλος οι ομιλητές μας. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 11. Ε, να καλωσορίσω λοιπόν τους ομιλητές μας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα σας δώσω το λόγο με τη σειρά που ήρθατε. Ελπίζω να μην ε, έχουμε, έχετε πρόβλημα. Ο κύριος ε, Ντομινίκα, ε, την, μετά η Ευρωπαϊκή ΕΑΤ, ο κύριος Αντζελόνι, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ρέιμοντ Ρόσπρειδ, εκτελεστικός διευθυντής της Εποπτείας Τραπεζών, ο κύριος Φράνκε από την ε, γερμανική Αρχή και ε, μετά από την, ε, το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης ο κύριος Σερένε Ρεπάζη. Ελπίζω ότι θα έχετε πάντοτε επίγνωση του χρόνου για να ολοκληρώνετε έγκαιρα τις ομιλίες σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας παρουσιάσω την πολωνική θέση σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση και ειδικότερα την πολωνική θέση σχετικά με την ενιαία τραπεζική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι η πρόταση της Κομισιόν που κατατέθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Να σας πω καταρχήν ότι η Πολωνία στηρίζει όλες τις δράσεις για την αύξηση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Την ανοικοδόμηση, την ε, ε, νέα εμπιστοσύνη στις αγορές και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων μεταξύ και της αρνητικής σχέσης μεταξύ δημοσίων, ε, δημοσίων οικονομικών και των τραπεζών. Ε, στην Πολωνία θέλουμε να αυξηθεί η τραπεζική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Κατά συνέπεια στηρίζουμε την ιδέα να δημιουργήσουμε μια τραπεζική ένωση. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό που συζητούμε τώρα, δηλαδή την ενιαία τραπεζική εποπτεία, είναι ένα μόνο από τα στοιχεία της ενότητας που ονομάζεται ε, τραπεζικό σύστημα ε, και είναι ένα στοιχείο για την εγγύηση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα. Στο μέλλον θα πρέπει να αποφύγουμε τα προβλήματα και τα λάθη που αντιμετωπίζουμε τώρα. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτές οι δράσεις δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Είναι μία μόνο δράση αυτή και μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα μόνο ε, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πώς μπορούμε να ε, επηρεάσουμε όλες τις συνιστώσεις που απαρτίζουν τον τραπεζικό τομέα. Φαίνεται ότι θα πρέπει να δούμε την Τραπεζική Ένωση όχι μόνο ως τραπεζική εποπτεία. Άρα λοιπόν χρειάζεται να συζητήσουμε για τη δημιουργία ενός καλύτερου συστήματος προστασίας και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου μηχανισμού, του μηχανισμού όπως λέγεται της εξυγίανσης των τραπεζών, που θα προστατεύει τις τράπεζες απέναντι στα οικονομικά προβλήματα. Τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συζητήσεων ήδη από τώρα και η Πολωνία πιστεύει ότι και τα τρία αυτά στοιχεία από κοινού μπορούν να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από μελλοντικά προβλήματα. Όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε πάλι ότι εμείς ως χώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη, Δεν είμαστε η χώρα που θα εφαρμοστούν άμεσα όλε αυτέ οι λύσει. Βεβαίω δεν αποθαρρύνουμε τη συζήτηση. Αντίθετα, τη θεωρούμε πολύ σημαντική και συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Θα έπρεπε να βρούμε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Να θυμόμαστε ένα πράγμα όμως, ιδιαίτερα όταν ε, εξελίσσουμε αυτό το σύστημα της ενιαίας εποπτείας. Όλες αυτές οι λύσεις ε, δεν μπορούν να μας ε, βάλουν στη διαδικασία ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς, την οποία αναπτύσσαμε στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα. Και οι προτάσεις που μπορούμε να δούμε τώρα μπορεί να οδηγήσουν στο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι άλλες τράπεζες. Αυτή η κατάσταση θα ήταν απαράδεκτη για την Πολωνία. Η τραπεζική... Ναι, λοιπόν, στην Τραπεζική Ένωση η τωρινή πρόταση δεν ανταποκρίνεται όμως ακριβώς στις προσδοκίες μας. Καταρχήν έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την συνεργασία με χώρες εκτός Ευρωζώνης η στενή συνεργασία, ο, ο μηχανισμός στενής συνεργασίας δεν δίνει ίσα δικαιώματα. Οι χώρες εκτός Ευρωζώνης έχουν λιγότερα δικαιώματα και περισσότερες υποχρεώσεις. Και βλέπουμε μάλιστα ότι για κάθε χώρα χωριστά οι κανόνες εξειδικεύονται στα πλαίσια της ενιαίας εποπτείας αν οι χώρες συμφωνήσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία και να ενταχθούν σε αυτή. Ε, πρέπει όλοι να έχουν ίδιους κανόνες, να υπόκεινται σε ίδιους κανόνες και όχι να ε, θεσπίζουμε ιδιαίτερους κανόνες για κάθε χώρα. Επίσης, πώς μπορεί να αποχωρήσει κανείς από αυτή τη δομή. Οι χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη και που θα είναι υπό την ενιαία εποπτεία δεν θα μπορούν να φεύγουν από τη διαδικασία αυτή γιατί αυτή η ε, οντότητα θα ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι τις επιμέρους τράπεζες. Αυτό ε, ενισχύει ακόμη περισσότερο την έλλειψη ισορροπία και δείχνει πως δεν είναι ίσα κατά τα δικαιώματα. Επίσης, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνουν σε τελευταία ανάλυση ότι η ισορροπία στην ΕΑΤ θα σπάσει γιατί η εκπροσώπηση θα ανατραπεί η ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διότι ε, θα εκφράζονται τα συμφέροντα των χωρών ε, υποδοχής και οι χώρες καταγωγής θα υπόκεινται σε άλλους κανόνες ισορροπίας. Δηλαδή θα υπάρχει ε, η δυνατότητα, οι αποφάσεις ε, της ΕΑΤ να αναφέρονται άμεσα και να ισχύουν για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα, θα δια, χρησιμοποιεί ένα φίλτρο για τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες χώρες δεν θα είναι απόλυτα υποχρεωμένες να ε, ε, ακολουθούν τους κανόνες. Είμαστε λοιπόν υπέρ της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά έχουμε πρόβλημα με κάποιες τεχνικές λύσεις της Κομισιόν και είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε για τις λύσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρώ μέσω στον Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η απόφαση του 2008 να αφήσουμε στα κράτη-μέλη και στις κυβερνήσεις τους όλη την ευθύνη για το θέμα του bailout μας οδήγησε τελικά σε μια χρηματοδότηση που είχε επιπτώσει στην πραγματική οικονομία. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήταν σωστό αυτό που είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του Χωσέ Γκαρσία Μαγάλιο και της Ελίζα Φερέιρα. Και βλέπουμε ότι σήμερα είναι επίγον να ξαναγυρίσουμε σε μια κανονική λειτουργία των αγορών. Βλέπουμε εδώ ότι η ταχύτητα δεν είναι αντίθετη με την ποιότητα. Και βλέπουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής με εξαιρετική ταχύτητα κάνει πολύ σωστές προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία με πολύ συγκεκριμένες ε, εξουσίες για την Ευρωζώνη. Αυτή η εποπτεία θα μπορεί βεβαίως εν μέρη να επιστρέψει στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα για κάποιε ιδιαίτερότητε των τοπικών αγορών. Εδώ υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλεία, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να επαφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό όσον αφορά την εξυγίανση. Αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Η διαχείριση για την επίλυση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας δείχνει ότι θα πρέπει η αναδιάρθρωση των τραπεζών να αποτελέσει προτεραιότητα κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα όπως ο μηχανισμός εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, EBA, καθώς και το θέμα της λήψης αποφάσεων και της ψήφου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία τελικά, εάν εφαρμοστεί, θα απαιτήσει σχεδόν ομοφωνία, κάτι που αποτελεί εμπόδιο. Προτείνουμε λοιπόν μια νέα πρόταση, ένα νέο μηχανισμό για τη λήψη αποφάσεων που θα λαμβάνει υπόψη ένα άλλο σύστημα και όχι την εκπροσώπηση των κρατών και κυβερνήσεων. Βλέπουμε ότι εδώ το θέμα είναι η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και όχι η σωστή εκπροσώπηση των εκπροσώπων των κρατών. Μία ψηφοφορία βάσει του συστήματος της πλειοψηφίας, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, σαφώς και θα πρέπει εδώ να προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα. Η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να μπορέσει... Αντρέα, προ... πάρα πολύ γρήγορα, διαβάζεις μάλλον πάρα πολύ γρήγορα, μπορείς να διαβάζεις λίγο πιο ναι, με ζητώ συγγνώμη, αλλά μου είπατε πέντε λεφτά. Έχω πολλά να πω. Εντάξει, θα τα πω πιο αργά. Να κάνω ό,τι μπορεί, Κάνω ό,τι μπορεί για να μπορούν να σε μεταφράσουν και οι διερμηνεί. Η Τραπεζική Ένωση τελικά θα πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά το ρυθμιστικό και αποπτικό πλαίσιο. Πολύ σημαντική πρόθεση έχει γίνει βάσει των απαιτήσεων για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τα πρότυπα που έχει προετοιμάσει η EBA, η Ευρωπαϊκή Αποπτική Αρχή. Χρειάζεται όμως εδώ να υπάρξει ένα σημαντικό επίπεδο για τη διακριτική ευχέρεια των κρατών. Σε σημαντικού τομεί τη ρύθμιση των τραπεζών, ιδιαίτερα όσον αφορά τι απαιτήσει σε κεφάλαιο, υπάρχουν ακόμα σημαντικέ πρόοδοι που πρέπει να γίνουν. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική ε, μεθοδολογία από τη μία χώρα στην άλλη. Πολλέ φορέ, δηλαδή ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες, βλέπουμε όμω ότι η εποπτεία μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση αποτελεί μια ευκαιρία να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα που εμπεριέχει το παρόν σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερη εναρμόνιση, ένα πιο ενιαίο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει σαφής ανάγκη για το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να γίνει πιο ενιαίο ιδιαίτερα όσον αφορά το βασικό κεφάλαιο και τις βασικές κεφαλικές ανάγκες. Η εποπτεία επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί εν ώψη των μαθημάτων που απορρέουν από αυτήν την κρίση. Ένα εγχειρίδιο για την σωστή διεκπαιρέωση αυτής της αποστολής είναι κάτι που θα χρειαστεί και θα πρέπει να συζητηθεί από όλους τους Εμπλεκόμενο σε αυτήν την εποπτεία. Δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση ένα εκτενέστατο εγχειρίδιο, αντίθετα θα πρέπει να αναλυθούν οι διάφοροι μέθοδοι εργασίες, να αξιολογηθεί η πολιτική των τραπεζών για την αξιολόγηση του κινδύνου και βεβαίως να υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, εποπτικής αντίδρασης. Ένα κοινό πλαίσιο για όλους αυτούς που θα ασκήσουν την εποπτεία, έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή στον εποπτικό μηχανισμό. Ένα εγχειρίδιο το οποίο θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να βοηθήσει να προσαρμοστεί η εποπτική πρακτική στις διαφορετικές πρακτικές των χρηματαγορών, στην αλλαγή η οποία είναι πολλές φορές ταχύτατη θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά την αξιολόγηση ε, των ε, κακών πρακτικών, των καταχρηστικών πρακτικών και των παραβιάσεων του ευρωπαϊκού νόμου, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Νομίζω ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας των περασμένων ετών, θα αλλάξει άσκηση της εποπτείας για τα επόμενα χρόνια, πάντα σε σχέση βεβαίως με το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε μια κρόαση πριν από δύο εβδομάδες εδώ, νομίζω σας ανέφερα τις σκέψεις μου για αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ, ο Ιγνάσιο. Thank you, Madam Chair. I'm, I'm very... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και είμαι πολύ ευτυχής και ε, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που με καλέσατε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω το κείμενο που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο ανταποκρίνεται πλήρως στι απαιτήσει που εξέφρασε η Ευρωζώνη τον Ιούνιο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την επικαιρότητα. Πρόκειται για ένα πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα βασικό ε, ε, στήριγμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ε, σε μια ολοκληρωμένη ζώνη η συλλογική λογοδοσία και εποπτεία είναι, συλλογική ευθύνη. Ε, τα τελευταία χρόνια και πρόσφατα στην υποπίεση έχει δημιουργηθεί μία δυσκολία όσον αφορά τη σταθερότητα και έχει αποδυναμώσει τον χρηματοπιστωτικό μας ε, τομέα και ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Υποβαθμίζει επίσης και υπονομεύει τις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης. Ο νέος μηχανισμός ε, μέσα σε αυτή την ε, ε, εικόνα θα πρέπει να εξασφαλίσει την συνεπή εποπτεία στην Ευρωζώνη και πέρα από αυτήν, καθώς και να αντιμετωπίσει το συστημικό κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί σε πολύ ολοκληρωμένους ζώνες να επηρεάσει για ε, την ε, μακροοικονομική σταθερότητα. Ο ενιαίος υπόπτης θα πρέπει άμεσα να ενεργεί και έγκαιρα απέναντι ε, στα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέψει έναν ορίζοντα νομισματική, χρηματοπιστωτική κατακαιρματισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση και νέο νόμισμα κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι επηρεάζεται και η ενιαία νομισματική πολιτική γραφώ σύντομα σε κάποιες ιδιαιτερότητες της πρότασης της ε, Κομισιόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα την εκτιμήσει λεπτομερώς σε την επίσημη γνωμοδότηση όπως απέτησε το Συμβούλιο και όπως απαιτείται από τη συνθήκη. Όμως ορισμένα στοιχεία είναι ήδη σαφή, ειδικά όσον αφορά τον ε, επιμερισμό που ανέφεραν οι δύο εισηγητές στην αρχή. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην εποπτική ευθύνη και στην, νομισματική, ε, ε, στην ευθύνη για την νομισματική πολιτική. Η Κομισιόν προτείνει αυτό να φτιαχτεί μέσω ενός εποπτικού συμβουλίου που θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων. Ε, το Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να μεριμνεί για τη διάκριση των δύο αυτών ε, τομέων υπάρχει καλή βάση για να εφαρμοστεί η αρχή αυτή της διάκρισης, ανεξαρτησία και η λογοδοσία θα πρέπει ένας ισχυρός υπόπτης να μπορεί να σταθεί σε κάθε πίεση ιδιωτικών και ειδικών συμφερόντων. Ε, Προλαμβάνονται ισχυρές διατάξεις ως προς αυτό, αλλά η εξαρτησία δεν μπορεί να είναι ισορροπημένη με ε, την αντίστοιχη λογοδεσία. Η πρόταση της Κομισιόν θεσπίζει τη λογοδεσία και τι αναφορέ για το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωγκρουπ. Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι η εποπτεία μπορεί να έχει και δημοσιονομικέ επιπτώσει. Ο νομοθέτη πρέπει να αποφασίσει το συγκεκριμένο περίγραμμα του πλαισίου για τη λογοδεσία. Και όπω ο πρόεδρο Δράγκη δήλωσε μόλι χθε, Είμαστε έτοιμοι να συμμορφωθούμε προ υψηλέ προδιαγραφέ λογοδεσία για τα επιπλέον αυτά καθήκοντα σε πλήρη συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτον, αποκέντρωση. Ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί ως ε, σύστημα που θα φροντίζει για την εμπειρογνωμοσύνη όλων των εθνικών εποπτών και ταυτόχρονα προσφέροντας ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει στενή σχέση με τις διάφορες κρατικές εποπτικές αρχές αλλά και ε, ισοτιμία μεταξύ του. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συλλέξει μεγάλη εμπειρία συνεργασίας με τι εθνικέ αρχές, κυρίως τι κεντρικές εθνικές τράπεζες, σε διαφορετικούς αλλά συγκρίσιμους τομεί. Τέταρτον, καθολικότητα. Έχουμε ε, μέσα στην πρόταση της Κομισιόν πολύ ισχυρές εποπτικές ε, εξουσίες ε, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ε, για τα μικρο και μάκρο ε, μέσα πρόβλεψης ε, ε, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στρέβλωσης που μπορεί να υπονομεύσουν την ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως αυτή η πρόταση είναι απόλυτα συμβατή με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ρόλος της EBA θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστός μέσω ενός ενιαίου κανον, ε, κα, κανονισμού και θα πρέπει να γίνεται υποπτία σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ε, EBA. Έχω εξάλλου συνεργαστεί επί μακρόν με τον Αντρέα και τους συναδέλφους του και είμαι βέβαιος πως η συνεργασία μας θα είναι εξαιρετική προς το συμφέρον της Ευρώπης. Πέμπτον, άνοιγμα. Ε, ε, καλωσορίζουμε την πρόταση των κρατών μελών να συνεργαστούν στενότερα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να είναι μέλη του υποπτικού μηχανισμού. Ε, η συμμετοχή των κρατών μελών θα πρέπει να διερευνηθεί όσο γίνεται περισσότερο μέσα στο νομικό πλαίσιο της συνθήκης και του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα πρέπει να αναλυθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τέταρτον, συγχρονισμός και επικαιρότητα προτείνεται ένα χρονοδιάγραμμα ε, πολύ φιλόδοξο, το οποίο όμως είναι εφικτό. Θα πρέπει να μπορέσει να υπάρξει μια σταδιακή είσοδο στο νέο σύστημα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο κανονισμός του Συμβουλίου να εγκριθεί όσο γίνεται πιο ε, σύντομα, γιατί διαφορετικά θα καθυστερήσει η προετοιμασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξεμεταλλευτεί την συμπληρωματικότητα και να αποφύγει την επικάλυψη. Έχει ήδη σημειωθεί πρόοδο σε ένα επικοδομητικό κλίμα. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Η έναρξη ισχύω του κανονισμού την 1η Πρώτου του 2013 θα διευκολύνει τη δημιουργία του Εποπτικού Συμβουλίου και την πρόσβαση στι πληροφορίε των τραπεζών των Ευρωζώνη, ώστε να υπάρξει ομαλή ε, και σταδιακή κίνηση του συστήματος. Χρειάζονται ωστόσο και άλλοι, άλλα στηρίγματα, κοινό σύστημα για την, ε, ε, για την εξαγορά και η διάλυση τραπεζών Ε, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αν υπάρχουν νομικές ε, και πολιτικές δυσκολίες. Οι αποτυχημένες τράπεζες που έχουν κάνει πτώχευση θα πρέπει να διαλύονται με συγκεκριμένο τρόπο χωρίς περιορισμού των εθνικών ε, εντολών. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά επόμενα βήματα. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνετε εδώ στην δίκησή μας πολλή δουλειά ξεπερνάτε το χρόνο και θα φύγω εκτός ελέγχου. Στη συνέχεια ο κύριος Ράιμοντ ε, Ρόζελεν. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση. Είναι τιμή μου ε, ε, που επιλέξατε εμένα για να εκπροσωπήσω την προοπτική του εθνικού επόπτη. Καταρχάς υποστηρίζω την έννοια ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και δεσμεύομαι να συνεισφέρω στην αποτελεσματική του δημιουργία και λειτουργία. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, στους οποίους η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να έχουμε καλά αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι ε, μπορεί και να καθυστερήσουμε και να μην ξεκινήσουμε τις εργασίες μας τον Ιανουάριο της 1η Ιανουαρίου του 2013 κάποιες διαδικασίες θα περάσουν από τις εθνικές εποπτικές αρχές ε, στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά ε, στην καιρό κρίση στην εποπτεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε το χρόνο μα και να σκεφτούμε γιατί έχουν αναλυφθεί οι δράσει. Οι προτάσει που συζητώνται δεν αφορούν ε, το να διορθώσουμε κάτι το οποίο είναι ε, σπασμένο. Ε, εγώ θεωρώ ότι η τραπεζική εποπτεία θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά η παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ε, ένας φαύλος κύκλος αρνητικός μεταξύ των ε, κρατών και των ασθενών τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως προϋπόθεση για να στηρίξουμε τις τράπεζες με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχάς, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ ελκυστική η διαδικασία της επέκτασης του πεδίου εφαρμογή της ε, εποπτικής αρχής ε, σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι σαφέ και δεν υπάρχει καμία εμφυσιμία. Στην ουσία όμω στην πράξη είναι αδύνατο για την άμεση εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επεκταθεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να λαμβάνονται πληροφορίε να αναλύονται και να λαμβάνονται αποφάσει. Η επιτυχής εποπτεία ε, δημιουργείται με ε, τακτικό διάλογο μεταξύ των τραπεζών που υπόκειται τον έλεγχο και καλή κατανόηση των τοπικών αγορών. Δεν νομίζω λοιπόν ε, ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο ότι θα, θα τον κάνει πολύ καλύτερα τον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Το πιο ρεαλιστικό θα ήταν να γίνει επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της, ε, ε, του εποπτικού συστήματος ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα εποπτεύουν συστομικά τις μεγαλύτερες τράπεζες και οι εθνικές εποπτικές αρχές θα είναι αυτές οι οποίες θα εποπτάζουν τις μικρότερες τράπεζες. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση της επιμερισμένης ευθύνη, θεωρώ ότι το βάρος του εποπτικού έργου ε, των ευρωπαϊκών σημαντικών τραπεζών θα πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά θα πρέπει να υπάρχει καθημερινή δέσμευση με τι τράπεζε, να κατανοήσουμε τι συναλλαγέ του, ε, να γίνεται ανάλυση των πληροφοριών και όλα αυτά είναι πολύ έντονα για να μπορέσουν να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μόνον, παρά ε, το γεγονό ότι μπορεί να πρόκειται για ένα πολύ μικρό αριθμό τραπεζών. Θα πρέπει να γίνονται όλα με βαθιά γνώση ταυτόχρονα και των τοπικών αγορών. Για παράδειγμα, η εποπτεία τη Deutsche Bank θα είναι ατελή ε, χωρί την ε, εποπτεία και τη θηγατρική της της ε, Postbank που είναι ένα σημαντικό παράγοντα στη γερμανική αγορά. Και φυσικά θα πρέπει να κατανοήσει πολύ καλά την τοπική αγορά για να εποπτεύει την Deutsche Bank. Επίσης θα πρέπει ε, οι επόπτες ε, να αναλαμβάνουν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλαμβάνει και αποφάσεις εποπτείας ναι. ε, και ορισμένες φορές θα πρέπει να φροντίζει για την υποχρεωτική εφαρμογή ή και κάποιες κυρώσεις για να μπορέσει να σπάσει ο φαύλος κύκλος αυτός. και αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από μία, πρέπει μάλλον να γίνει συγγνώμη, από μία αρχή, είτε αυτή θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Οι τράπεζες δεν θα γνωρίζουν όμως ε, πού μπορούν να προσφύγουν για να αναθεωρηθεί μια τέτοια απόφαση. Οι βασικές αρχές της Βασιλείας ε, απαιτούν, ε, να υπάρχει ένα κατάλληλο και ε, σταθερό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και αυτό σημαίνει ότι οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Εποπτικών Φορέων θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς στον κανονισμό του Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή υπάρξει σαφήνεια για τον κατάλληλο επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και κατανομή του έργου, το επόμενο βήμα θα είναι να υπάρχει ένας κοινό στόχος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική εποπτείας με περισσότερες λεπτομέρειες και θα πρέπει να γίνει καταμερισμός σε προγράμματα εποπτείας και επιθεωρήσεων για τις τράπεζες και τους τραπεζικούς ομίλους. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε μια κοινή εργαλειοθήκη, κυρίως να υπάρχει μια συμφωνία για το πώς γίνεται η εποπτεία. Και η στρατηγική και αυτή η κοινή εργαλειοθήκη θα πρέπει να υπάρχουν πριν μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι ο εποπτικό μηχανισμό είναι σε πλήρη λειτουργία. Και αυτό θα χρειαστεί χρόνο και δεδομένου ότι βιώνουμε και χαλοπού καιρού ε, θα πρέπει να ε, προηγηθεί ε, το κατάλληλο προηγούμενο και όχι το κατεπήγον, ο κατεπήγον χαρακτήρας του συγκεκριμένου γεγονότος. Για να μπορέσουμε να μην δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική πορεία, ένα πιο ρεαλιστικό χάρτη πορείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν ε, περάσω στον τελευταίο μιλητής, ομιλητή, θα ήθελα τα μέλη που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις ή να κάνουν κάποια παρατήρηση να μας το πούνε και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα τα μέλη και μετά να δώσουμε το λόγο στο πάνελ για να απαντήσει γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή mm. μας. Ευχαριστώ. Good morning, Madam Chairwoman Bowles. Καλημέρα σας ε, κυρία Πρόεδρε Μπόλς, αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής, ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Ευχαριστώ που με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση για την ε, εποπτεία των τραπεζών. Είμαι εδώ ως νομικός ε, ε, εμπειρογνώμων και θα ήθελα να παρουσιάσω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, η επιλογή της νομικής βάσης του άρθρου 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης και το θέμα των εκτελεστικών εξουσιών. Δεύτερον, το τίμημα που θα καταβληθεί για αυτή την επιλογή που είναι η επισφαλής συμμετοχή των κρατών μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Τρίτον, η αρχή τη δημοκρατίας όπως προστατεύεται από τις συνθήκες της Ένωση και τα συντάγματα των κρατών μελών και το πεδίο εφαρμογή ε, της εγγύηση ανεξαρτησίας τη ΕΚΤ. Τέταρτον, το θέμα των εναλλακτικών που γυρίζει γύρω από το ερώτημα ποιος φοβάται τον Μερώνη. Οι τωρινέ προτάσεις ε, του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, δίνουν εποπτικά καθήκοντα στην ΕΚΤΕ με βάση τη νομική βάση του άρθρο 127 παράγραφο 6 της συνθήκη για τη Λειτουργία την Ένωση. Ο βασικός λόγος για την επιλογή αυτής της νομικής ε, βάσης ήταν το γεγονός ότι το πρωτογενέ δίκαιο δίδει εκτελεστικέ εξουσίε στην ΕΚΤ με βάση το... Επειδή ήδη προβλέπει το πρωτογενές δίκαιο τέτοιου είδους εκτελεστικές εξουσίες δεν χρειάζεται η ΕΚΤ ε, κατεξουσιοδότηση εκτελεστικέ πράξει που θα έθεταν τα γνωστά θέματα για την απόφαση Μερώνη. Το τίμημα για τις ε, περιόρισες εκτελεστικέ εξουσίες είναι η επισφαλή συμμετοχή των κρατών μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη στον ενίο εποπτικό μηχανισμό. Ο λόγος είναι το άρθρο 139 της συνθήκη, που αποκλεί την εφαρμογή κάποιων συνθήκων ε, προβλέψεων τη συνθήκη στα λεγόμενα κράτη-μέλη με εξαίρεση που είναι τα μικρά, τα κράτη-μέλη που δεν είναι στην, ε, ε, ζώνη του ευρώ. Το άρθρο 139 προβλέπει ότι οι εκτελεστικές εξουσίες, το άρθρο 132 της ΕΚΤ ε, και η συμμετοχή των οργάνων λήψη αποφάσεων της ΕΚΤ δεν εφαρμόζονται στις χώρες που δεν είναι, ε, που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Μία συμμετοχή των κρατών μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη στα όργανα λήψη αποφάσεων της ΕΚΤ όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί από αυτή τη συμφωνία του μηχανισμού στενής συνεργασίας. Ε, τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων γιατί Ήδη η λήψη αποφάσεων στο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπεται. Υπάρχουν δύο όργανα λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Το να υπάρξει κι άλλο όργανο μέσα στην ΕΚΤ για να, που να έχει δικαιώματα λήψη αποφάσεων, αυτό θα παραβίαζε τι συνθήκε και δεν μπορεί να αλλάξει χωρί αλλαγή τη συνθήκη. Έτσι λοιπόν το τίμημα που θα ε, πληρώσουμε για την επιλογή τη ΕΚΤ ω βασικού παίχτη στον ενίο μηχανισμό ε, είναι ότι τα κράτη-μέλη που δεν είναι στην Ευρωζώνη δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων μέσα στην ΕΚΤ. Ακόμα και το νέο λεγόμενο εποπτικό συμβούλιο υποτίθεται που θα ε, σχεδιάζει και θα εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ δεν μπορεί να υποχρεώσει νομικά το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση που μπορεί να ε, σχεδιάσει. Η αρχή της δημοκρατίας και της ε, τραπεζικής υποπτίας. Εδώ έχουμε την αρχή της δημοκρατίας ε, που περιορίζεται ε, σε σχέση με μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από το Γερμανικό Σύνταγμα και τον, ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ασκεί συγκεκριμένα καθήκοντα που αφορούν την τραπεζική υποπτία δημιουργεί όμως ένα κενό. Η τραπεζική υποπτία είναι ιδιαίτερα πολιτικό θέμα και οι εποπτικές αποφάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στα άτομα. Ε, έλλειψη δημοκρατική λογοδοσία είναι ιδιαίτερα προβληματική σε σχέση με την αρχή τη δημοκρατία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι αντίθετα με αυτό που ισχυρίζονται πολύ συχνά, η εγγύηση ανεξαρτησία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζεται στην τραπεζική εποπτεία. Αυτό ε, προκύπτει πρώτον από τη διατύπωση τη εγγύηση για την ανεξαρτησία στο άρθρο 130 τη συνθήκη, που ε, αφορά μόνο καθήκοντα και υποχρεώσει που έχει η ΕΚΤ ε, βάσει των συνθήκων και του καταστατικού ε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο στόχος του άρθρου 130 είναι να ε, διασφαλίσει την ανεξαρτησία στις σε σχέση με την νομισματική πολιτική της Ένωσης. Ε, όμως ε, η, εποπτεία δεν έχει να κάνει με την νομισματική ε, τόσο πολύ. Γι' αυτό η ρήτρα για την ανεξαρτησία δεν θα ήταν α, εμπόδιο στην άμεση λογοδοσία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού του ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο ή κάποια ειδικά δικαιώματα για ε, έρευνες. Ε, τέλος, ε, για κάποιους το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για την επισφαλή συμμετοχή των ε, κρατών που δεν είναι στην Ευρωζώνη είναι πολύ ψηλό. Για άλλους η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την νομισματική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύεται από την τραπεζική εποπτεία. Αυτό φέρνει στην επιφάνεια το θέμα διαφορετικής θεσμικής ρύθμισης και διαφορετικής νομικής βάσης. Όποτε αρχίζει η συζήτηση για το θέμα αυτό, θυμάμαι το πιο σοβάται τον κακό λύκο από τα τρία μικρά τα τρία γουρουνάκια και ποιος φοβάται το Μερόνι. Αυτή η απόφαση του 58 ήθελε να προλάβει την εκτελεστική εξουσία από το να δώσει εκτελεστικές εξουσίες σε όργανα εκτός ε, πολιτικού ή νομικού ελέγχου. Τώρα έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια ε, ολοκλήρωση του δικαίου και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Καταρχήν με τη συνθήκη της Λισαβόνας η δράση για ακύρωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, επεκτάθηκε σε ε, ε, πράξεις σωμάτων, οργάνων και φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομική προστασία είναι δεδομένη και δεύτερον, εις ό,τι αφορά τις, τους ελέγχους και τις ισορροπίες, η εκτελεστική δεν μπορεί να δώσει περισσότερες εξουσίες από, από αυτές που έχει, που ήταν η περίπτωση Μερώνη. Ο νομοθέτης λοιπόν έχει ελευθερία να ε, δώσει εκτελεστικές εξουσίες και διακριτικές ε, εξουσίες στο βαθμό που ε, ο επαρκής έλεγχος αυτών των εξουσιών μπορεί να διασφαλίζεται. εδώ θα πρέπει να συμβουλευτούμε το άρθρο 290 της συνθήκης. Επίσης, σε αυτά τα πλαίσια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, θέτει σαφή όρια σε μια τέτοια ε, ανάθεση εξουσιών ε, διατάξεις που για να υιοθετηθούν απαιτούν πολιτικές αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της νομοθετικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να εξουσιοδοτούνται. Για να συνοψίσω, κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ, ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα πρέπει καταρχήν να είναι πιο δημοκρατικά, να, να ε, ε, προβλέπει δημοκρατική λογοδοσία, λογοδοσία και δεύτερον να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερα κράτη-μέλη για να ε, είναι διασφαλισμένη η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες λύσεις εκτός από το προτινόμενο άρθρο ως νομική βάση. Ε, νομίζω ότι θα ε, πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για να επιληθούν όλα τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον ένας από τους εισηγητές έχει ερωτήσεις. Ίσως ήταν πιο λογικό να ακούσουμε πρώτα τα ερωτήσεις από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές και έπειτα αντί να κάνουν μια σύνοψη στο τέλος οι εισηγητές να, ακούσω, να υποβάλουν τι ερωτήσει που θα έχουν εκείνη την ώρα αφού θα έχουν ακούσει και τι τις ερωτήσεις των υπολείπων. Όλοι χρειάζεται να πάρουν το λόγο. Οπότε προσπαθώ να βρω τώρα ποιοι είναι οι σκιώδεις εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Νίτρας πρώτος. Ε, E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω κάποια σχόλια καταρχήν. Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Πάση. Ρε Πάση, συγγνώμη. Ε, όταν ακούμε ε, μάλλον ε, εκτιμώ τα επιχειρήματα, αλλά έχω κάποιε αντιρρήσει όσον αφορά τι χώρε εκτό Ευρωζώνης. Ε, κατανοώ ότι η συνθήκη είναι έτσι, αλλά αυτό το άρθρο αναφέρει κάποια ειδικά καθήκοντα όσον αφορά την εποπτεία. Όχι όλα τα καθήκοντα ή ολόκληρο το συνολικό σύστημα. Βλέπω λοιπόν να υπάρχει εδώ κάποια διαφορά. Ε, από τη μια πλευρά δηλαδή αναφέρεται το άρθρο αυτό όταν μιλάτε για την ε, αδυναμία των χωρών εκτός Ευρωζώνης να συμμετέχουν. Από την άλλη πιστεύω πως το άρθρο αυτό δεν αναφέρεται στο σύνολο της εποπτείας αλλά σε κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένα άλλο ε, αίτημα που έχω είναι αν μπορείτε να σχολιάσετε και τώρα αναφέρομαι στην συμβολή του κυρίου Ενρία. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς καθημερινά συνεργάζεστε με τα θεσμικά, του θεσμούς, ε, τους τραπεζικούς ε, σε εθνικό επίπεδο. Από ό,τι, από είπατε, κατάλαβα ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως και συγχρονισμένα, αλλά είπατε επίσης πως η ΕΚΤ είναι σε καλύτερα προετοιμασμένη για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να αρχίσει να παίζει τον ρόλο ενός ε, μιας τραπεζικής εποπτικής αρχής την 1η Ιανουαρίου για όλα τα τραπεζικά θεσμικά όργανα στην Ευρώπη. Όπως ήδη απόθηκε είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, θα πρέπει να γνωρίζετε την αγορά πάρα πολύ καλά, να γνωρίζετε ποια είναι η η αλληλεπίδραση, η συνεργασία ε, μεταξύ όλων αυτών. Αν δείτε όλες τις αγορές από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, οι αγορές διαφέρουν πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε ότι η προθεσμία, η ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου. Αλλά εγώ πραγματικά ανησυχώ και φαντάζομαι πως πολλοί έχουν τις ίδιες αμφιβολίες. Αν δείτε ας πούμε τους ε, όσους έχουν υπηρεία από την εποπτεία τραπεζών ε, θα έχουν, έχουν τις ίδιες αμφιβολίες. Ο Υπουργός Ντομένικα ανέφερε κάποια στοιχεία. Πώς σας φαίνεται αυτή η ημερομηνία, πώς πρέπει να καταλάβουμε αυτή την ημερομηνία. Είναι πραγματική, είναι ρεαλιστική, είναι εφικτή ή είναι ε, προϊόν φαντασίας. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν σα είπα από την αρχή πόσο χρόνο έχετε, αλλά επειδή ε, άρχισα να μετράω τα λεπτά, παρακαλώ να περιοριστείτε στα τρία λεπτά για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε τι απαντήσει των εμπειρογνωμόνων. Να σα πω ποιου έχω στη λίστα μου. Έχουμε κατά ομάδες I've got Gunnar Hockmark and then Marion Tyson at the end. From the S&D, I've got Elisa Ferreira, Peter Simon, Roberto Galtieri and Antolin Sanchez Prosedo. From LD, I have Sylvie Goulard and Olli Schmidt. ECR, I don't have anybody. Από την ECR δεν έχω κανέναν για την ώρα και από τους πράσινους τον Φίλιπ Λάμπερτ και μετά τον Σβέν βέβαια. Η Ελίζα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω και συμφωνώ με πολλούς ομιλητές που είπαν ότι πρόκειται για μια ευκαιρία. Πρόκειται για μια ευκαιρία μοναδική που θα έχουμε για να κάνουμε κάτι. Ωστόσο καταλαβαίνω κάποια από τα ερωτήματα τα οποία ήδη τέθηκαν πιο συγκεκριμένα. Μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα ανάμεσα στα εθνικές εποπτικές αρχές και το νέο ρόλο της ΕΚΤ μέσω της αποσαφήνισης των ορίων που, ορίζον, που χορηγούνται στο στους εθνικούς, στο Εθνικό Όργανο Εποπτείας και μπαίνοντας σε πιο λεπτομερή προσέγγιση για το σε ποιο βαθμό το σώμα των, το εποπτικό θα παίξει κεντρικό ρόλο για τη λήψη απόφασης από πλευράς ΕΚΤ. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση διότι η ΕΚΤ έχει κάποιες ε, ισχυρές ε, εξουσίες ε, παρέμβασης ως επόπτης που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα για ορισμένες χώρες όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ακόμα και εντός της Ευρωζώνης. Οπότε μπορούμε να λύσουμε μήπως κάποια από αυτά τα δύσκολα προβλήματα αποσαφηνίζοντας σε πιο λεπτομερώς πώς ε, μπορούμε να μοιραστούμε και πώς ε, ο ενιαίος επόπτης ε, θα μπορεί να εποπτεύει κατανοώντας όμως τα εθνικά συμφέροντα και τις εθνικές ευαισθησίες θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα δικαίωμα έφεση, α πούμε, για σε μια απόφαση τη ΕΚΤ. Αν η ΕΚΤ αποφασίσει κάτι που είναι πολύ ε, ριζοσπαστικό, πώ θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι η σχέση ανάμεσα στην φάση εποπτείας και τη φάση διάλυσης, ή εξαγορά τράπεζας μιλήσατε για ένα κοινό εγχειρίδιο πρακτικής. Όχι μόνο όμως για υποπτικά θέματα, θα πρέπει να είναι αυτό να ισχύει και για περιπτώσεις εξαγοράς ή, ή διάλυσης τράπεζας ώστε στη μεταβατική αυτή φάση να υπάρχει μια κοινοτική ε, ε, προσέγγιση και σχετικές διατάξεις και στις δύο περιπτώσεις. Πώς βλέπετε λοιπόν τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που εποπτεύει, ενώ όταν έρχεται η φάση διάλυσης η εξαγοράς θα έχει τις πληροφορίες ταυτόχρονα στη διάθεσή της για να ε, ε, ε, ελέγξει τις αρχές εξαγοράς ή διάλυσης της τράπεζας. Έπειτα, βλέπετε να υπάρχει ε, δυνατότητα για ένα κοινό, ε, κοινό πλαίσιο διάλυσης τραπεζών μέσα στην Ευρωζώνη τουλάχιστον. Έπειτα, βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα ο ρόλος της ΕΚΤ να διευρυνθεί σε όλες σε όλα τα μέλη της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δυνατότητα ε, opt-out για τις χώρες. Λίζα, συγγνώμη, δεν, δεν βάλαμε μπροστά το χρονόμετρο. Γλίτωσε σε 1,5 λεπτό. Έχουμε και διαπραγματεύσει που πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε εδώ. Ξεχάσαμε το χρονόμετρο. Εντάξει, εντάξει, πείτε μου πότε τελειώνει ο χρόνος. Α, συγγνώμη και νόμιζα ότι τα είχα πάει τόσο καλά, τα είχα πει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ε, Δεδομένης τώρα της κατανομής ανάμεσα στις ομάδες, να ακούσουμε ακόμα έναν από τους σοσιαλιστές, τον Πίτερ Σίμων. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις στον κύριο Αντζελόνη από την Εκτε. Η πρώτη αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφος, από την, συνάδελφός σας από την Μπάφιν. Είπε πολύ συγκεκριμένα γιατί πιστεύει ότι ο έλεγχος μέσω των ε, μικρότερων τραπεζών θα πρέπει να παραμείνει στις εθνικές εποπτικές αρχές. Εσείς είσαστε πιο συντηρητικός. Μιλήσατε για την ε, συνεργασία των δύο και είπατε ότι θέλετε να αποφύγετε επικαλύψεις. Εσείς συμφωνείτε με αυτά που είπε ο συνάδελφός σας από την Μπάφιν και αν όχι, πού θα ε, κάνατε κριτική και πού θα αντιπαρατεθείτε σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Μπάφιν. Μια δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην εξυγίανση. Resolution. Λέτε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε ε, όσο γίνεται περισσότερο να ε, κρατήσουμε το φορολογούμενο μακριά από αυτές τις εξυγιάνσεις. Βλέπω τις προτάσεις της Κομισιόν όμως που λένε 1% ε, ε, ε, κάλυψη από τις καταθέσεις για το resolution. Θα πρέπει αυτά να είναι ως προϋποθέσεις. Οπότε πάμε σε 78 δις στην Ευρώπη. Η τελευταία κρίση στήχησε 400 δις. Αυτά ήταν οι δαπάνες άμεσης ανακεφαλαιοποίησης. Εσείς με τις προτάσεις της Κομισιόν και, και το Bail-in έχετε να αντιπαραθέσετε δικές σας προτάσεις ούτως ώστε να γλιτώσει από την ε, επώδυνη συμμετοχή στο μέλλον ο φορολογούμενος. Ευχαριστώ. Σιλβί. Καταρχήν, επειδή ήμουν μία από τις εισηγήτριες, δεν πρόκειται για μία και μοναδική ευκαιρία Ήδη είμαστε στη δεύτερη προσπάθεια, άρα πραγματικά ας είμαστε πιο μετριοπαθείς. Θα δούμε τι θα προτείνουμε και τι θα δεχθούν κατόπιν τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω στον εκπρόσωπο του Μπάφιν. Πολύ συμπαθητικό αυτό που μας είπατε. Πολύ συμπαθητικό. Όλοι θέλουν ευρωπαϊκή εποπτεία υπό όρους υπό όρους, ποιους όρους ο εθνικός επόπτης θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε από αυτό το σύστημα. Δεν λέω ότι όλα πρέπει να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση. Αλλά το θέμα είναι, έχουμε αποφασίσει να είμαστε σοβαροί, ναι ή όχι. Είδατε τι είπε το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο, ότι πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τις τράπεζες κτλ. Και μία ερώτηση για τον κύριο Ρεπάση όσον αφορά την δημοκρατία, το δημοκρατικό έλεγχο. Εγώ δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη σοβαρά μιλούν για λογοδοσία. Όλα τα μηνύματα που βλέπουμε μας δείχνουν ότι δεν είναι και πολύ σοβαρή όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας, accountability. Ας αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα πολιτικά ορθά που ακούμε όσον αφορά τη δημοκρατία, όσον αφορά τη λογοδοσία και τις υποχρεώσεις. Αλλά η ερώτηση είναι πολύ σοβαρή και δεν έχω ακόμα ακούσει την απάντηση. Πώς μπορεί κανείς να έχει ένα τέτοιο σύστημα λογοδοσίας και εδώ στρέφομαι και προς τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης, οι οποίοι θέλουν να εκπροσωπούνται στο εποπτικό ε, συμβούλιο, στο όργανο που θα ασκήσει την εποπτεία. Και αναρωτιέμαι, είτε πρέπει να επιλέξουμε άλλη νομική βάση, Αλλιώς θα πρέπει να αποφασίσουμε ή παραμένουμε στο άρθρο 127.6 και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η βάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σημαίνει πρόβλημα με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και πρόβλημα λογοδοσίας είτε θα δώσουμε άλλου είδους προτεραιότητες και σε αυτή την περίπτωση δεν παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παραμένουμε σε ένα άλλο όργανο το οποίο ενδεχομένως θα στεγάζεται στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας φιλώ και τους πέντε και πείτε μας, είσαστε πέντε κύριοι που θα μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Πρόεδρος, πριν προχωρήσω στον Φιλίπ Λαμπέρ, θα ήθελα να πω τους ε, εμπειρογνώμονες ότι έχετε μόνο τρία λεπτά για να απαντήσετε. Σας το λέω γιατί μπορείτε βεβαίως να στείλετε και γραπτές απαντήσεις. Με μεγάλη χαρά θα τις δεχτούμε. Γιατί ξέρω ότι είναι αδύνατον μέσα σε τρία λεπτά να απαντήσετε σε όλα αυτά που σας ε, τέθηκαν σαν ερωτήματα. Ο Φιλίπ. Ευχαριστώ. Το ερώτημά μου, το ερώτημά μου απευθύνεται στον εκπρόσωπο της Μπαφίν. Α, συγγνώμη, ο Ζων Πολ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι εδώ προετοιμάζουμε μία ακρόαση. Δίνουμε πέντε λεπτά στον ε, μιλητή, τρία λεπτά να απαντήσει. Και εντωμεταξύ, εμείς ακούμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και δεν έχουμε απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την παρουσία των εμπειρογνωμόνων. Εντάξει, ήρθαν στις Βρυξέλλες, ίσως για να δουν και τα αξιοθέατα των Βρυξελών, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ας τους δώσουμε 8 λεπτά, αυτό προτείνω, για να μας απαντήσουν για ένα θέμα που απασχολεί όλους στην Ευρώπη, που είναι η κρίση και η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Επαναλαμβάνω, δεν έχω ερώτηση, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που ήδη έχω πει, ότι η οργάνωση αυτών των ακροάσεων Χολένη. Πρόεδρος. Ζαν Πολ, γνωρίζεις πολύ καλά από τους συντονιστές ότι τα προβλήματα που έχουμε στο χρονοδιάγραμμα και στα σχέδια η δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για την Επιτροπή μας γιατί δεν επιτρέπεται. Λυπούμε, ε, συμμερίζομαι το πρόβλημά σου. Εγώ σκοπεύω να μην χρησιμοποιήσω τα τρία μου λεπτά. Η ερώτησή μου είναι προ τον κύριο Μποντχόβερ. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και να προσέξουμε, μην διαλέξουμε λάθο αρχιτεκτονική. Όμω έχω κάποια προβλήματα με αυτό που είπατε. Καταρχήν, μιλήσατε για το γεγονό ότι ο επόπτη πρέπει να ξέρει την αγορά και άρα πρέπει να είναι κοντά. Είναι γνώμη μου ότι η υπερβολική η ε, συνάφεια βλάπτει. Ε, οπότε μπορεί να δείξει δηλαδή ο επόπτης επίκαια. τι θα τώρα, η Deutsche Sparkassen είναι συστημική ή όχι απέναντι στην αντίστοιχη Ισπανική που κάνει την ίδια δουλειά. Η εντύπωση που έχω εγώ, ακούγοντας τον Μπάφεν και άλλους από τη Γερμανία, είναι ότι η πειθαρχία είναι καλή για τους άλλους, αλλά αν εμείς μπορούμε να την αποφύγουμε θα ήταν καλύτερα. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν σε αυτά. Μάλκομ, για όσους διαμαρτύρονται για τη σειρά με την οποία τους δίνω το λόγο, δεν ε, είχαμε κατσιδιά, είχαμε κατά ομάδες τις καταλαγούς και προσπαθώ να κάνω μια κυκλική ε, επιλογή. Μου το ζητήσατε σε προηγούμενες ακροάσεις, ο Γκούναρντ είναι επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα, αντιμετωπίζουμε νέες ενώσεις, νέα σχήματα, πολιτική ένωση, δημοσιονομική ένωση και διάφορες άλλες ενώσεις που έχουμε φεύρει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση που υπάρχει και η οποία αντιμετωπίζει και δημοσιονομικά θέματα και πολιτικά και οικονομικά. Και ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολούν είναι βεβαίως αυτό το κοινό εγχειρίδιο κανόνων. Και αυτό σαφώς είναι και στην καρδιά αυτών που συζητούμε. Αφορά την εγγύηση των καταθέσεων, τις απαιτήσει σε κεφάλαιο και τις λύσεις για εξυγίανση και καθάριση τραπεζών. Και πιστεύω ότι πολλές φορές θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο Και θεωρούμε ότι ακριβώς και μόνο το γεγονός ότι είναι καινούριο θα είναι και καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας, αλλά θα ήθελα να ζητήσω πολλούς εμπειρογνώμονες να μας παρουσιάσουν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τον κατακαιρματισμό των χρηματαγορών, δημιουργώντας νέους θεσμούς, κινδυνεύουμε να φύγουμε μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Και βεβαίως όλοι θέλουμε εποπτεία Όλοι θα θέλαμε να υπάρξει εποπτεία, ιδιαίτερα που να ξεπερνάει προβλήματα τα οποία καλύπτουν όλη την επικράτεια της Ευρώπης. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει ο κατακαιρματισμός, ότι υπάρχει μια εποπτεία με επικαλύψεις και ενδεχομένως θα μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις γιατί πρόκειται για πολύ καλού εμπειρογνώμονε που έχουμε σήμερα εδώ. Πρόεδρο. Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο Αντολίν Σάντσε Πρεσέντο, ο Όλι Σμιτ και στη συνέχεια ο κύριο Γκίκολτ. Ρομπέρτο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση και να θέσω και μία ερώτηση προς τον κύριο Ρεπασί ε, για το νομικό του επιχείρημα, διότι το βρήκα πολύ πιστικό με έπεισε όλη η ομιλία με την εξαίρεση του σημείου αυτού της αντίφασης μεταξύ τη δυνατότητα να εκχωρούμε την εποπτεία ε, στον ε, ε, εποπτικό φορέα και τα δικαιώματα ψήφου στον στο μηχανισμό διαχείρισης. Ο εποπτικός φορέας είναι το Εποπτικό Συμβούλιο που βάσει συνθήκης δεν έχει μέλη εκτός Ευρωζώνης. Ίσως όμως αυτή η αντίφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί εάν έχουμε την αρχή της κυριαρχίας της συνθήκης σε σχέση με το πρωτόκολλο. Διότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αντίφαση βάσει του άρθρου 10 με βάση το άρθρο 10 σημείο 1 του πρωτοκόλλου. Και δεδομένου ότι αφορού, συζητούμε νέα καθήκοντα, τα οποία είναι καθήκοντα τα οποία δεν καλύπτονται από το παρόν καταστατικό, Υπάρχουν επιπλέον καθήκοντα λοιπόν που εκχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω μια ειδική νομοθετική διαδικασία, η οποία έχει ένα καθεστώ το οποίο συγγενεύει με την αλλαγή τη συνθήκη. Επομένως έχουμε κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 7,6 του καταστατικού. Πρόκειται λοιπόν για μια συγκεκριμένη απόφαση που σχετίζεται με τον εποπτικό μηχανισμό και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι ε, διοικητές των ε, τραπεζών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην εξαιρούνται από την όλη διαδικασία. Είτε μέσω μιας ε, μορφής συνδικαλιστικής συμφωνίας, μιας μορφής δημοσιονομικού συμφώνου και να ψηφίζουν και οι άλλοι λαμβάν, σαν να λαμβάνεται υπόψη η ψήφο τους ή ως ένα επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, είστε βέβαιοι ότι ε, δεδομένου ότι συζητάμε νέα καθήκοντα, τα οποία δεν καλύπτονται από το καταστατικό, δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε αυτή την αρχή της κυριαρχίας υπόψη και να υπάρχει μια παρέκκληση για τους διοικητές των τραπεζών εκτός Ευρωζώνης που θα μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που δεν είναι εκτελεστικές μόνο, αλλά είναι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντολίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι όταν συζητάμε την κρίση, ως λύση για την κρίση ε, δώσαμε στο παρελθόν μία λύση που μου θυμίζει αυτά που κάναμε στο 16ο αιώνα που συζητούσαμε τα θέματα της θρησκείας. Υπήρχε συνθήκη του Αψβούργου ε, και λέγαμε ε, τι πρέπει να κάνουμε με τη θρησκεία. Εφαρμόζει, εφαρμόζεται η θρησκεία του κυρίαρχου κράτους για τους πολίτες. Και εδώ ουσιαστικά εφαρμόζουμε την κυρίαρχη αξία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήγηκε η ώρα να καταλήξουμε σε μια διαφορετική λύση. Η εποπτική αρχή, ο μηχανισμός εποπτείας ε, εδώ ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη με βάση την νομισματική πολιτική. Διότι η νομισματική πολιτική είναι το κόστος της καταναλωτικής πίστης, της ε, πίστης ε, των ενυπόθηκων δανείων, των δανείων για τις επιχειρήσεις και όχι ποιος είναι ο κυρίαρχος σε αυτή την περίπτωση. Η άποψή μου λοιπόν είναι... Καταρχάς να σταθώ στον κύριο Ντομινίκ. Εάν το βασικό μας θέμα είναι η νομισματική πολιτική, θα μπορούσαμε να ε, δούμε τι γίνεται μόνο με δύο κράτη-μέλη, που είναι τα κράτη-μέλη που έχουν παρέκκληση, γιατί όλα τα υπόλοιπα ε, θα ήταν σε μεταβατικό καθεστώς ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μέλλον στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια μεταβατική λύση. Θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο για να συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Για τα δύο κράτη τα οποία είναι εκτό είναι προφανέ ότι δεν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε αυτό το μηχανισμό, διότι θέλουν να έχουν ξεχωριστό νόμισμα και επομένως θα πρέπει να αναζητήσουμε μεταβατικές λύσεις. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένας ε, κάποιος μηχανισμός συνεργασίας για τις άλλες δύο. Επίσης, η διαφορά είναι όντως ε, να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια οικονομική και νομισματική ένωση. Ποιος ε, είναι αυτό ο οποίο θα διακρίνει αυτό το στοιχείο εποπτεία από την υπόλοιπη εποπτεία που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία ερώτηση τώρα. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώ μπορεί κάποιο να βρίσκεται και εντό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάποιο μηχανισμό και ταυτόχρονα να είναι και ξεχωριστό. Ε, έχετε κάποια πρόταση, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Ε, να έχουμε αυστηρά νομισματική πολιτική από τη μία και ε, ε, χρηματοπιστωτική υποπτία από την άλλη. Ε, θα πρέπει αυτά να τα συνδυάσουμε και με την πραγματική οικονομία και την νομισματική πολιτική ταυτόχρονα. Κύριε Αντζελώνη. Η αρχή ότι όλοι οι υποπτικοί φορεί θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στον νέο υποπτικό μηχανισμό διότι υπάρχουν ε, και συστημικές ευρωπαϊκές τράπεζες και εγχώριες τράπεζε. Ε, πώς θα πρέπει να διαμορφώσουμε το μηχανισμό ώστε να δούμε πώς έχουμε άμεση εποπτεία, πώς μπορούμε να έχουμε ένα πιο κεντρικό μηχανισμό και ένα πιο άμεσο σε τοπικό επίπεδο. Και στον κύριο Ρόσελερ από τον Μπάφιν. Στο τέλος αναφερθήκατε σε ρεαλισμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ρεαλισμός είναι ότι είναι βιώσιμη η κατάσταση όσο έχει τώρα. Μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές διατηρώντας το status quo ή θα πρέπει να καθορίσουμε άλλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, διότι αυξάνονται οι κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ταυτόχρονα αρχίζουμε να μεταφέρουμε προβλήματα ε, ιδιωτικού εξωτερικού ε, χρέους σε ε, ευρωπαϊκό χρέος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις πολιτικής φύσεως στον κύριο Ρέσλερ. Μιλάτε για ε, συμφόρηση. Μετά τις 28-29 Ιουνίου δεν υπήρξε ένα τέτοιο πρόβλημα που καθυστέρησε, που, θα, που καθυστέρησε τις αποφάσεις ε, δεν είναι μια μεγάλη συμφόρηση γιατί είναι σοβαρές οι πολιτικές αποφάσεις. Είχαμε 18-19 συνεδριάσεις, ο καθένας τις ερμήνευε διαφορετικά όταν γύριζε στην πατρίδα του και τώρα προβλέπεται και άλλη συνεδρίαση. Μου φαίνεται ότι ακόμα και για τη Γερμανία και για το δικό σας ίδρυμα ίσως θα ήταν κάτι επικίνδυνο. Για τον Πολωνό Υφυπουργό Οικονομικών εσείς πόσο σκληρά θα παίξετε αν οι προϋποθέσεις που θέτετε δεν υπάρξουν. Πόσο σκληροί θα είστε. Θα μπλοκάρετε τη συνέχεια ή θα πείτε θα συνεχιστεί η Ευρωζώνη και θα υφίσταται χωρίς εμάς. Αυτές είναι οι πολιτικές μου ερωτήσεις. Πόσο σκληρή είναι η Πολωνία. Ευχαριστώ. Πίσω στους ε, εισηγητές μας. Παρακαλώ μην υπερβείτε τα τρία λεπτά ή δυνατόν. Η Μάριαν. Ε, ε, Ευχαριστώ, θα είμαι... Έχω, έχω. Θα είμαι σύντομη. Είπαμε για τη στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αναφέρομαι στην Πολωνία. Χρειάζεται μια εξήγηση εδώ. Αν θέλει μια ε, χώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη να συμμετάσχει ε, μπορεί να γίνει μια παρασκευαστική δουλειά μέχρι να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Γιατί να θέλουν να φύγουν, βέβαια, ίσως παρουσιάσουν λόγους. Εκτός από αυτά, ο Πολωνός υπουργό είπε ότι δεν μπορούν να γίνονται χωριστές ε, διαπραγματεύσεις για τη στενή συνεργασία. Ίσως ε, και οι άλλοι εμπειρογνώμονες ε, έχουν να μας πούν πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να υπάρξει μια γενική προσέγγιση με τα κριτηρία της Κοπενχάγης ως βάση για παράδειγμα και να συμφωνήσουμε για το ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν παράλληλα με τα προηγούμενα της Κοπενχάγης. Τώρα για το αν θέλει κανείς να προσχωρήσει ή όχι στο, στην διαδικασία αυτή. Ο κύριος Φερέιρα το ανέφερε αυτό πιο πριν. Είναι δυνατόν, πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες, να αντιστραφεί το σύστημα και να υπάρχει opt-in δυνατότητα να προσχωρεί κανείς και μετά να αποχωρεί opt-out. Ε, επίσης ε, δεν είναι μόνο ε, ενιαίο βιβλίο αλλά ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Θα ήθελα να πω στην ε, στην ε, ΕΚΤ. Τι θα είναι αυτό, θα είναι κάτι που θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τέλος μια γρήγορη ερώτηση στο νομικό ε, εμπειρογνώμονα για την απόφαση Μερώνη. Λέτε ότι δεν μπορεί οι εκτελεστικές εξουσίες να δίνονται σε άλλον από την ΕΚΤ. Ε, λέτε ότι δεν μπορούν δηλαδή να δίδονται ε, στην ΕΚΤ θα πρέπει να βρούμε άλλη εναλλακτική. Κάποιος πρέπει να δει τα νομικά θέματα γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς σήμερα ακούσαμε μία νομική άποψη, αλλά δεν είμαι βεβαία ότι είναι η μόνη. Μπορεί να είναι η βασική, η επικρατούσα, αλλά υπάρχουν κι άλλες νομικές απόψεις. Οπότε κάποια στιγμή οι πολιτικοί θα πρέπει να βρουν τη λύση σε τελευταία ανάλυση. Υπάρχουν πάντως και άλλες νομικές σχολές σκέψης. Ευχαριστώ Μάριανο Σβέν. Πολύ σύντομα, δεν θέλω να βαρεθείτε ακούγοντας να επαναλαμβάνονται οι ερωτήσεις. Θέλω να επαναλάβω κάτι που έμεινε ανοιχτό, θεωρώ, από την αρχή. Απευθύνομαι κυρίως στον εκπρόσωπο της ΕΚΤ. Μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι η λογοδοσία και η υποβολή εκθέσεων στο, είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωζώνη αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι για το opt-in, πώς θα υποβάλλετε έκθεση στην Ευρωζώνη. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεύτερον, ε, για το, την ειλικρίνεια ή το άνοιγμα λέτε ότι πρέπει να γίνεται προσεκτική ανάλυση του εφικτού στα πλαίσια του κανονισμού ΕΚΤ. Ε, θέλω να μου πείτε εσείς τι είναι δυνατόν και εφικτό σε σχέση με τις ε, δυνατότητες λήψης αποφάσεων των χωρών που προσχωρούν στα πλαίσια της ΕΚΤ. Θέλω να μου πείτε η θέση δική σας ποια είναι. Τέλος, ε, στον Ρενέρα Ρεπάζη, εσείς μας λέτε δηλαδή ότι τα όρια για τη συμπερίληψη των χωρών οπτήν δεν μπορούν να ξεπεραστούν στα πλαίσια των συνθήκων. Δηλαδή υπάρχει άλλος τρόπος για να υπάρξει μια πραγματική ε, εποπτεία στην Τραπεζική Ένωση στο πλαίσιο των συνθήκων και ποια θα είναι η νομική βάση για να ισχύσουν όλα αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τα μέλη. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δώσουμε πάλι το λόγο στους ομιλητές μας. Πέντε λεπτά στον καθένα, καλός χρόνος είναι αυτός. Πάλι με την ίδια σειρά έχει νόημα αυτό. Ε, θα επιλέξετε τα πιο ζουμερά και μετά θα ε, πείτε στα άλλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Τα βασικά θέματα για την Πολωνία που αφορούν την όλη αυτή τη συζήτηση, ώστε να έχουμε δηλαδή έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, είναι τα εξής. Καταρχά, ένα νέο σύστημα, ε, νέο μηχανισμό εποπτείας δεν θα πρέπει να δημιουργήσει κι άλλου περαιτέρω κατακαιρματισμού μεταξύ ευρωπαϊκών τραπεζών και τραπεζών εν γέννη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ε, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, αν είναι εντό ευρωζώνης ή εκτός ευρωζώνης. Θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασία για τον τραπεζικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πριν από ένα-δύο χρόνια αποφασίσαμε να υπάρχει ενιαία τραπεζική αγορά. Δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε διαφοροποίηση επειδή κάποιε τράπεζε είναι από την Ευρωζώνη και κάποιε τράπεζε είναι εκτό Ευρωζώνη και τη χάνουν διαφορετική προστασία. Δεύτερο στοιχείο. Η μεταφορά, εκχώρηση των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από ε, εκχώρηση ευθυνών για τις ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ιδίως ε, τις χρηματοοικονομικές ευθύνες. Είναι απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα, ιδίως για χώρες εκτός Ευρωζώνης, να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες τους επιβάλλονται και ταυτόχρονα η όλη ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές να, απόκειται σε αυτούς. Και εμείς από εκεί και πέρα να πρέπει να υποστούμε τις οικονομικές συνέπειες για τις συγκεκριμένες αποφάσεις, ενώ δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποβάλουμε ένσταση για τις αποφάσεις αυτές. Κατόπιν, στο συγκεκριμένο στάδιο, για να είναι κανεί επιτυχή, δεδομένου ότι είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι ε, συστηματικά ε, σημαντικέ τράπεζε, ιδίω αυτέ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή εποπτεία για τι τράπεζε αυτέ, ιδίω λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ε, ισορροπία μεταξύ των χωρών κρατών, χωρών μελών συγγνώμη, που τις ε, φιλοξενούν. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί καταλήλως ακόμα σε ε, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, το ε, πού ε, είναι η κεντρική τράπεζα και ποια χώρα τη φιλοξενεί δεν έχει ακόμα διευθετηθεί. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα, να βρούμε τη δέουσα ισορροπία για την εποπτεία των χωρών μελών που φιλοξενούν ή έχουν την έδρα τους οι, οι τράπεζες. Επίσης, ακούστηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, μεν, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί είναι πολύ κακή η εμπειρία μας από το 2008-2009. Υπήρχε ένα διάστημα ε, ανεξέλεγκτης αύξησης ε, των εγγυήσεων των καταθέσεων ε, στα κράτη-μέλη και όλοι γνωρίζουμε τι συνέπειες είχαν αυτά. Μέσα σε ελάχιστες ώρες η γειτονική τραπεζική τομή σε γειτονικές χώρες ε, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Η, τεράστια μεταφορά καταθέσεων από τη μία χώρα στην άλλη μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια στο τραπεζικό τομέα σε διάφορε χώρε. Γνωρίζουμε τι έγινε στη Σλοβενία και σε άλλε χώρε λόγω αποφάσεων που έλαβαν οι γειτονικέ του χώρε. Πλέον λοιπόν, όταν θα ετοιμάσουμε αυτό το νέο σύστημα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ε, διασπάσουμε αυτή την ισορροπία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μπορεί να δημιουργηθεί ανάλογη κατάσταση και Αφενός με να έχουμε ένα προστατευμένο ε, σύστημα το οποίο την χάνει υποπτίας εντός της Ευρωζώνης και οι χώρες εκτός ε, να μείνουν ε, στο έρμο των αποφάσεών τους. Τώρα, για την ερώτησή σας το πόσο σκληρή είναι η Πολωνία. Καταρχάς, δεν είναι θέμα του πόσο σκληροί είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ αποφασισμένοι να διαπραγματευτούμε μια καλή λύση για όλη την Ευρώπη διότι πραγματικά ε, σκεφτόμαστε σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη στο μέλλον ε, και αυτή τη στιγμή διανύουμε μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν θα συζητηθεί το νέο σύστημα, όπως έγινε και στο παρελθόν, όλο το ευρωπαϊκό σύστημα δημιουργήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη τη στιγμή, παρά το γεγονό ότι ε, κάποιοι εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη και κάποιοι όχι. Όλοι είχαν τα ίδια δικαιώματα στη διάρκεια των συζητήσεων και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα. Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό για μας αυτή τη στιγμή, τότε απλώς θα αναβάλουμε την ένταξή μας ε, στο σύστημα, στον ενίο επεπτικό φορέα, μέχρι τη στιγμή που η Πολωνία θα ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση, να έχουμε απλώ υποχρεώσεις και να μην υπάρχει καμία επιρροή από πλευράς μας στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you. Well, quite a lot of... Uh, πάρα πολύ σημαντικά θέματα και θα προσπαθήσω να επιλέξω μεταξύ αυτών τα πιο σημαντικά. Πρώτον, ταχύτητα. Κάνατε μια ερώτηση για την ταχύτητα και πόσο καλά προετοιασμένη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ θα ήθελα να πω εδώ ότι καταρχήν το ερώτημα είναι γιατί είναι επίγον. Γιατί, διότι σήμερα χρησιμοποιούμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων γιατί ακόμα δεν λειτουργεί το άλλο σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν να ενδυναμωθεί το σύστημα ευρωπαϊκού ελέγχου, ευρωπαϊκής εποπτείας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει και εμείς το ίδιο. Αλλά θα είναι πολύ σημαντικό το συντομότερο δυνατόν να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα καλύπτεται η χρησιμοποίηση ευρωπαϊκού χρήματος με τη δυνατότητα πραγματικού ελέγχου όσον αφορά την καλή χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Γι' αυτό και θα πρέπει η Επιτροπή να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν αυτή την επευθεία ιδιαίτερα για τις τράπεζες αυτές που έχουν επωφεληθεί από τα χρήματα αυτά, από τη χρηματοδότηση αυτή. Μιλήσατε για, την, για τον κατακαιρματισμό. Ναι, βεβαίως, αυτό υπάρχει. Και υπάρχουν πολλές εποπτικές διαδικασίες ήδη. Αυτό δεν είναι αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με, το ευρωπαϊ... με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά αυτό ουσιαστικά επιδεινώνει και ενισχύει τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Και τελικά το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η ενιαία αγορά. Επίσης, μικρές τράπεζες και μεγάλες τράπεζες. Για μένα το σημαντικό σημείο είναι ότι αν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, ότι κάποιες τράπεζες δηλαδή εξαιρούνται από την κάλυψη αυτής της ευρωπαϊκής εποπτείας, από το φάσμα της ευρωπαϊκής εποπτείας, σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουμε να βρεθούμε στον εξή ε, κίνδυνο. Κάποιες τράπεζες να έχουν δίκτυο ασφαλείας και κάποιες όχι. Αυτή τη στιγμή η ανησυχία των χρηματαγορών εστιάζεται στην ισχύ αυτού του δικτύου ασφαλείας που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε περισσότερη σταθερότητα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αυξήσουμε τους κινδύνους σε κάποια σημεία. Τρίτο σημείο, όσον αφορά την εξυγίανση, εκαθάριση. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικά τα όργανα εδώ, είναι πολύ σημαντικά τα διάφορα σώματα και η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Η συλλογική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία λήψη αποφάσεων γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτά τα συλλογικά όργανα να μην περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη λήψη αποφάσεων ο μηχανισμός θα πρέπει να απλουστεύσει αυτή τη διαδικασία. Και όσον αφορά την εξυγίανση, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Πρόκειται για μια διαδικασία δύο φάσεων. Στην πιο μακροπρόθεσμη φάση θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προσέγγιση της, των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα αυτό και ίσως αυτό θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε μια αρχή στην Ευρώπη και μια διαδικασία όσον αφορά αυτή την αρχή που είναι αρμόδια για την εξυγίανση και την εκαθάριση και πιστεύω ότι η εποπτική αρχή θα πρέπει να εξελιχθεί προς αυτή την απόφαση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ε, Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τα εκεί κατά την άποψή μου. Τώρα, το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, καταμερισμός των ευθυνών και των εξουσιών. Ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προετοιμάσει ένα εγχειρίδιο για όλες τους επόπτες. Το κύριο συστατικό αυτού του εγχειριδίου θα πρέπει να εστιάζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου στην εκτίμηση του κινδύνου, με ποιο τρόπο γίνεται, με σκοπό βεβαίως να παραμείνει η ενιαία αγορά και να λειτουργεί. Υπό την αιγίδα πάντως της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να ειδωθεί αυτό το εγχειρίδιο. Ο Ιγνάτσιο. Πρόεδρε, ήταν πολύ ζουμέρε όλε οι ερωτήσει για να το πω όπω το είπατε κι εσεί. Εγώ έχω σημειώσει μόλι έξι, ομαδοποιώντα τα σχόλια που έγιναν. Καταρχήν, η κατανόηση των τοπικών αγορών. Δηλαδή, πρέπει κανεί να διατηρήσει ένα σχετικό βαθμό εγκύτητα στην πραγματικότητα των τοπικών αγορών και να βρίσκεται κοντά στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα στι χώρε όπου υπάρχει μέγα τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπω. Γερμανία και Ιταλία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό και η απάντησή μου μοιάζει με αυτή του κυρίου Λαμπέρα, ότι δηλαδή υπάρχει πλεονέκτημα όσον αφορά τη γνώση, την εγκύτητα, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος, αν κανείς είναι εξαιρετικά κοντά στην τοπική πραγματικότητα, να παραβλέψει κάποια στοιχεία ε, ομοιομορφίας, ε, ισοτιμίας, ε, ισότιμου πεδίου που πρέπει να επικρατήσει σε ένα τομέα, σε μια περιοχή μάλλον όπως η Ευρωζώνη και πέρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα τον είπα είναι αξιδάμαστο προς πολλούς βαθμού και το ένα, ο ένα τομέα είναι η διάλυση, η εξαγορά επιχειρήσεων. Αλλά μια πτυχή σχετίζεται με αυτό το σημείο περισσότερο. όπως ξέρετε, έχουν δύο επίπεδα εποπτείας, δηλαδή είναι ο πολιτιακός και τοπικός και ο άλλος είναι για την, σε εθνικό επίπεδο για τις εθνικές τράπεζες και αποδείχθηκε από έρευνες σχετικά με τις τράπεζες ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση ανάμεσα στα δύο στρώματα, ότι δηλαδή η κρατική είναι πιο επίκη από ότι η ομοσπονδιακή. Αυτό είναι, ένα, είναι ήδη αναγνωρισμένο μέσα στις ε, σχετικές έρευνες. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εγκύτητα και το ε, αμεροληψία. Επίσης τώρα, δεν θα πρέπει κανείς να συγχαίει τα, τα κονδύλια για την κρίση με τα κονδύλια για διάλυση τραπεζών, γιατί για τα κονδύλια για την κρίση συμπεριλαμβάνουν και τα κονδύλια για την ε, διάσωση, το bailout, ενώ για την ε, εκαθάριση η εξαγορά μιας τράπεζας ε, είναι πολύ μικρότερα τα ποσά συνήθως. Ε, ε, επαγγελματική μας περηφάνεια είναι να μπορούμε να καθαρίσουμε μια τράπεζα με μίνιμουμ αντίκτυπο στο τραπεζικό τομέα και χωρίς χρήση κονδυλίων. Καμία χρήση κονδυλίων ξεπληρώνουν έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της καθάρισης κάποιας τράπεζας. Ε, ελπίζω πως αυτό θα μπορούμε να το καταφέρουμε από τη στιγμή που θα έχουμε μία ενιαία αρχή εκαθάρισης για την Ευρώπη που όπως είπα στην εισήγησή μου πρέπει να είναι ένα από τα επόμενα βήματα. Τώρα, το, η χρήση του 1276 σαν νομικό ε, μέσο το Συμβούλιο αποφάσισε από αυτού και είναι και νομική αναγκαιότητα θα έλεγα γιατί η συνθήκη έχει προβλέψει το συγκεκριμένο μέσο για να επιτύχει το συγκεκριμένο ρόλο. Να παίξει το συγκεκριμένο ρόλο. Λοιπόν, απαραίτητο να δούμε αυτό το μέσο πριν να διερευνήσουμε άλλα. Εγώ το θεωρώ και ως ευκαιρία γιατί το 127.6 επιτρέπει να ληφθούν αποφάσεις και δίνονται αρμοδιότητες που έχει η ΕΚΤ. Ε, ο υπόπτης έτσι αποκτά πολύ ισχυρέ ε, αρμοδιότητες. Δεν είδαμε τι έχει συμβεί με τέτοιο χρήμα. Άστε να έχουμε έναν επόπτη, ο οποίος να είναι στη θέση να λάβει ε, αποφάσεις προς το συμφέρον της Ένωσης. Πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός, αυτό ήταν το ερώτημα του κ. Σάντζες Περέρα. Εγώ εξέτασα τις ε, διεθνείς αποδείξεις και βλέπουμε ότι ακόμα και εθνικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τίνει να υπάρχει περισσότερη συγκέντρωση στην κορυφή, σε οποιαδήποτε δομή. Είτε οι αποφάσεις είναι γενικιακά εφαρμοστές, δηλαδή εφαρμόζονται για όλες τις τράπεζες, είτε αναφέρονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις κάποια σημασίας βέβαια. Έχουμε αυτά τα δύο είδη δράσεις λοιπόν που εν γέννη τα βλέπουμε στο κέντρο. Στην... Είναι ένα κέντρο το Εποπτικό Συμβούλιο, αλλά συμπεριλαμβάνει και τους εθνικούς επόπτες. Και η απόφαση που αφορά περισσότερο την τοπική πραγματικότητα και δεν μπορούν, δεν μπορούν να εφαρμοστούν γενικά, μπορούν να αποκεντρωθούν με πλήρεις αμοιβέ ε, πληροφορίες σε όλες τις περιπτώσεις, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι. Αλλά η συγκεκριμένη δράση του επόπτη θα ληφθεί από την Εθνική Εποπτική Αρχή. Η κυρία Τίσεν και ο κύριος Γκίγκολντ, τελευταίες μου παρατηρήσεις. Εποπτικό εγχειρίδιο, Ανδρέα που απάντησε ήδη και συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι εγώ θεωρώ το εγχειρίδιο που μπορεί να πρέπει να προετοιμάσει ο επόπτης της ΕΚΤ ως πλήρως συμβατό και συνεπές με τα όσα θα συντάξει η Ευρωπαϊκή Εποπτική, Τραπεζική Αρχή που είναι εντολή της να συντάξει τέτοιο εγχειρίδιο εφόσον θα ισχύσει διάφορες πραγματικότητες μάλλον θα είναι γενικού επίπεδου αλλά θα, πρέπει, θα δούμε αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και για την προσκάνη της εσωτερικής οργάνωσης του συστήματος που βέβαια δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει σε την EBA. Ε, Πάντως θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των δύο. Τώρα, λογοδοσία του Eurogroup και δυνατότητα να επιτύχουμε ή όχι, τι είναι εφικτό και τι όχι. Ναι, το Eurogroup μπορεί να είναι μια αρχική δυνατότητα όπου καλύπτονται όλες οι χώρες της Ευρωζώνης και μετά θα ήταν σκόπιμο, μόλις καταστεί δυνατόν, και το λέω αυτό από την πλευρά της ΕΚΤΕ, Μόλις θα μπουν και άλλε χώρες και θα έχουν στενή συνεργασία μαζί μας, ναι βεβαίω. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η λογοδοσία εκεί και να συμπεριληφθούν και οι αρμόδιες αρχές από τις χώρες που συνεργάζονται στενά. όπου τι είναι και τι είναι δυνατόν και τι όχι. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά από νομικής άποψης δεν θεωρούμε πως είναι τόσο ακραίο αυτό και υπάρχουν διάφορες απόψεις, όπως είπε και η κυρία Τέισεν για την υπόθεση Μερώνη και άλλα. Λοιπόν, ε, εφόσον υπάρχει ευρεία χρήση του Εποπτικού Συμβουλίου, εντάξει, να πω δύο λόγια, να πω δύο λόγια. Όχι, σας προειδοποίησα για να κλείνετε. Εντάξει, 15, 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια τάση και υπάρχει ανάγκη για εξέβρεση της ε, καλύτερης δυνατής ε, λύσης σε συνδυασμό ανάμεσα στις δραστηριότητες και τις ευθύνες του Εποπτικού Συμβουλίου και το δυνατότητες ε, ευελιξίες που έχουμε για να διοργανώσουμε την διακυβέρνηση του Εποπτικού Συμβουλίου. Και σε αυτό το παζάρι, θα έλεγα, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο συνδυασμό, δίνοντας μια κεντρική θέση και στις χώρες που συνεργάζονται στενά, στο Εποπτικό Συμβούλιο μια επιλογή είναι βέβαια οι εξουσίες ε, ψήφου, η ψήφοι του καθενός και θα πρέπει να το δούμε από νομική άποψης και να λάβουμε υπόψη ότι θέλουμε το εποπτικό αυτό συμβούλιο να αναλάβει διάφορες σημαντικές δραστηριότητες. Αν υπάρχει αυτή η τάση, πρέπει να βρούμε την καλύτερη νομική λύση και αυτό το μελετάμε. Λυπάμαι που μακρηγόρησα. Ναι, τι να σας πω, παλιότερα ήμουνα πιο αποτελεσματική. Κοιτούσα με άγριο τρόπο τους ομιλητές και αυτό τους έκανε να σταματούν. Φαίνεται ότι δεν πιάνω πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά αυτά τα πολύ περίπλοκα ερωτήματα, επιτρέψτε μου να μιλήσω στα γερμανικά. Το ερώτημα του κατά πόσο εδώ υπάρχει η ανητική επίπτωση. Θα ήθελα να πω βεβαίω, εδώ πρέπει κάποιο να γνωρίζει τις τοπικές αγορές. Εννοείται. Εγώ παραδείγματο χάρη αν ε, πρέπει να ασκήσω εποπτικό έλεγχο στην Ιταλική αγορά, στο Ιταλικό τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να απευθυνθώ στους αρμόδιους, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και αν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εποπτεία υπέρ των τραπεζών, θα πρέπει αυτό να μπορεί να γίνει με πλήρη τρόπο. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν με γρήγορο τρόπο και απερίσκεπτα να μεταφέρουν όλο το τραπεζικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για εκατοντάδες, χιλιάδες αποφάσεις το χρόνο. Πώς μπορεί αυτό να το κάνει, να το διεκπαιρεώσει μόνη της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Και πραγματικά θα πρέπει να περιοριστούμε σε κάποιες μεγάλες τράπεζες όπου θα υπάρχει προστιθέμενη αξία ε, στο να διεκπεραιώνεται ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε όλες και όχι στις μικρότερες. Τώρα, το θέμα του ποιος είναι, ποιος μπαίνει στην κατηγορία συστημικών και ποιος όχι τραπεζών. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των τραπεζών, ένας μεγάλος, μια μεγάλη ομάδα τραπεζών που δεν μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Και το έχουμε συζητήσει αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να ταξινομήσει τις τράπεζες και αυτό πάντα έχοντας κατά νου τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. Πώς μπορεί κάποιος να καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο αυτών των τραπεζών. Και το θέμα είναι Εάν δεν καταφέρουμε να λάβουμε την απόφαση στην 1η Ιανουαρίου και ποιος θα ευθύνεται και ποιες θα είναι αρνητικέ συνέπειες, κατά την άποψή μου θα είναι πολύ χειρότερο να βρούμε μία μη καλή απόφαση και να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Γιατί εκεί αυτό που θα κάνουμε είναι θα αποσύρουμε τις αρμοδιότητες από τις εθνικές αρχές και δεν θα είμαστε σε θέση να καλύψουμε αυτήν την διαδικασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Ο κύριος Ζωραπασί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς να απαντήσω το ερώτημα της δυνατότητας του opt-in και του opt-out στο σχετικό άρθρο. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να περάσουμε σε ένα μοντέλο βάσει του 27-6 ε, σε μοντέλο opt-out. Το είπε και ο κύριος Αντζελόνη στην αρχική του παρέμβαση. Ο βασικός στόχος για την επιλογή της συγκεκριμένη νομικής βάσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εφαρμοστικές εξουσίες βάσει πρωτογενούς δικαίου, αλλά αυτές οι εφαρμοστικές εξουσίες βασίζονται στα κράτη της Ευρωζώνης και για τα κράτη μη Ευρωζώνης θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, εκτελεστικές εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει τέτοιες εκτελεστικές εξουσίες, επομένως η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του opt-in για να λέμε ότι η εθνική νομοθεσία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να προβλέψει τι ε, σχετικέ εκτελεστικέ εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χωρί αυτέ, δεν υπάρχει νόημα για την τραπεζική εποπτεία. Επομένως, ε, βάσει τη Συμφωνία Στενή Συνεργασία, ένα κρατό μέλο έχει τι απαραίτητε εκτελεστικέ εξουσίε σε εθνικό επίπεδο, ε, οι οποίε είναι απαραίτητε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Με βάση αυτού μπορούμε να πάμε λοιπόν στη δεύτερη παρατήρηση για την υπόθεση Μερώνη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καταρχάς γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των νομικών, ε, αυτό δεν θα έπρεπε να σας εκπλήξει. Λέμε πάντα ότι όταν υπάρχουν δύο νομικοί υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις. Ε, αυτό είναι κανόνας. Η υπόθεση Μερώνη λοιπόν δεν ισχύει για την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και γιατί δεν ισχύει. Ο κύριος Αντζελώνη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκτελεστικές εξουσίες που τους εκχωρούνται μέσω πρωτογενούς δικαίου από τις συνθήκες. Η υπόθεση Μερώνη για τις ε, κατεξουσιοδότηση ε, δεν ισχύει γιατί δεν υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση κατεξουσιοδότηση πράξης. Μπορεί κάποιο να πει ε, ότι υπάρχει ανάγκη εξουσιοδότηση πράξεων για τα κράτη εκτό Ευρωζώνη. Εδώ όμω το, 127, το 127 παράγραφο 6 αναφέρει διεξοδικά πώς μπορεί να εκχωρηθεί η δυνατότητα της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το Εθνικό Δίκαιο. Και επίσης, πώς μπορούν να διεξαχθούν αυτά τα καθήκοντα, με ρωτήσατε. Κατά την άποψή μου, η 127.6 προβλέπει κάτι το οποίο είναι δυνατό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μόνο μέσω αλλαγής της συνθήκης μπορούν να ε, ε, χωριθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με μία εξαίρεση την τραπεζική υποπτία και εδώ πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κατοίκοντα. Η συνθήκη όμως ε, δεν λέει ότι δεν μπορεί να ανατεθεί η τραπεζική υποπτία σε κάποιον άλλον φορέα, όπως για παράδειγμα την EBA ή κάποιον άλλο φορέα με νέα νομική βάση. Και εδώ έρχομαι ε, στην ερώτηση του κυρίου Γκίγκολτ. Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ξέρω ότι από πολιτική σκοπιά το να αλλάξουμε τελείως τη μέθοδό μας δεν είναι ότι πιο φρόνιμο. Επιτρέψτε μου όμως ε, ε, να πω κάτι για το θέμα αυτό θεωρώ ότι το άρθρο αυτό μας παρέχει νομική βάση για να ε, κάνουμε κάτι τέτοιο. Διότι, όπως σας είπα, το 127.6 ισχύει μόνο για, το, ε, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ το 352 ισχύει για οποιοδήποτε άλλο φορέα. Εγώ θεωρώ ότι κανονικά θα έπρεπε να το αναλάβει η EPA. Αλλά αν δεν θέλουμε να το δώσουμε στην EPA, το 352 μας δίνει την κατάλληλη νομική βάση για να δημιουργήσουμε ένα νέο φορέα που θα αναλάβει την εποπτεία και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη δυνατότητα opt-in και opt-out. Οι λύσεις opt-out βάσει του 352 μπορούν να εφαρμοστούν και επομένω μπορούν να χρησιμοποιούν βάσει του συγκεκριμένου άρθρο. Το άρθρο 352 επίσης προβλέπει και τη δυνατότητα ομοφωνίας ε, όπως και το 127.6 και επομένως δεν αλλάζει ο τρόπος λήψης απόφασης στο Συμβούλιο. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη διαφορά. Το 352 προβλέπει και σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το 127.6 ε, προβλέπει ε, μόνο απλώς τη γνωμοδότησή σας. Και αυτή είναι η μόνη υποβάθμιση που γίνεται στο Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης, διότι σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται συνένεση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε έναν εποπτικό φορέα στον οποίο όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα μπορούν να αποφασίσουν από κοινού για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα βάσει του 352. Το 352 βέβαια έχει κάποιους περιορισμούς, δεν είναι η τέλεια νομική βάσο, βάση, η δάλλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την είχε επιλέξει. Πρόκειται όμως για μια καλή εναλλακτική λύση. Να περάσω τώρα στο θέμα της αρχής της κυριαρχίας. Δεν νομίζω ότι η αρχή της κυριαρχίας θα δώσει λύση στο πρόβλημά μας, παρά το γεγονός ότι πολύ θα το επιθυμούσα. Σε σχετικό άρθρο της συνθήκης ε, λέγεται ότι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις ε, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και τα εποπτικά σώματα. Καθορίζεται λοιπόν σαφώς ποιοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν και επίσης λέγεται ότι τα πρωτόκαλα έχουν την ίδια αξία με τη συνθήκη και επομένω η αρχή της κυριαρχίας μπορεί να ισχύει μόνο όταν υπάρχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις ανάμεσα στις, ε, ε, σε δύο φορείς. Επομένως πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή λοιπόν, για να τροποποιήσουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και όπως είπα, αν θέλετε να υποβάλλετε και άλλα έγγραφα, θα είμαι θα... ιδιαίτερα ευγνώμονες. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ακρόαση, αφού αλλάξουμε εδώ τη σειρά μας. Okay, if you could see, take your seats, then I can see who's here. Καθίστε για να δούμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι εδώ. Okay. Thank, thank you very much to our panel. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Συγγνώμη που έπρεπε να σας ζητήσουμε να βγείτε και να συνεχίσουμε. Κλέψαμε μία ώρα από ένα πιο μεγάλο hearing για τις τράπεζες σε κρίση. Καθίστε λοιπόν. Αυτό ήταν το αρχικό ε, hearing και ευχαριστώ τον Γκούναρ που μας παραχώρησε κάποιο χρόνο που ήταν για την έκθεσή του. Τώρα θα μιλήσουμε λοιπόν για τις τράπεζες σε κρίση και θα δώσω το λόγο στον Γκούναρ Χόκμαρκ, τον εισηγητή, να κάνει προκαταρκτικές παρατηρήσεις και μετά θα περάσουμε στους τρεις ομιλητές, τον Μπο Λούντγκρεν, τον προκαθηγητή Γκούντερ Φρανκ και τον ε, πρόεδρο Κρίστιαν Κλάουζε. Και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές που απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας. Αυτό είναι ένα και σημαντικό κομμάτι από το ενίο εγχειρίδιο κανόνων και χρειάζονται συζητήσεις για να έχουμε τραπεζικό σύστημα δυναμικό και ασφαλές όσο γίνεται περισσότερο. Ας δούμε κάποια θέματα που καλό είναι ίσως να συζητηθούν στην ακρόαση αυτή. Θα ήθελα οι ομιλητές να τα καταπιαστούν τα προβλήματα αυτά για να αναδείξουν τα προβλήματα και την επίλυσή τους. Μια γενική παρατήρηση πρώτα. Συχνά στη συζήτηση λέμε ότι ελπίζουμε να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις. Όλοι βέβαια θα συμφωνούσαν με αυτό αλλά δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδομένο ότι γιατί ό,τι και να κάνουμε κρίσεις θα προκύπτουν, διάφορες κρίσεις ε, και μέσα από διάφορα πρίσματα ειδωμένες. Το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε ή όχι κρίσεις στο μέλλον. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτές και πώς θα τις αντιμετωπίζουμε όταν έρχονται. Και, ίσως το πιο σημαντικό, πώς θα βγαίνουμε από τις κρίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Πρέπει λοιπόν να τα δεχτούμε αυτά ως πραγματικότητα. Όσο πιο έτοιμοι είμαστε, όσο πιο αυτοσχεδιάζουμε σε μια κρίση, και βέβαια εδώ αυτή η οδηγία σκοπό έχει να μας ε, κάνει έτοιμους, ε, αυτά είναι θέματα που πρέπει να βλέπουμε και θα μας τα πούν οι ομιλητές. Ένα άλλο θέμα είναι το εξής, ότι ε, οι κρίσεις διαφέρουν. Μπορεί να είναι μία τράπεζα σε κρίση. Και στο άλλο άκρο μπορεί να έχουμε τραπεζική κρίση, συστημική, γενικευμένη. Νομίζω ότι η φύση και ο χαρακτήρας αυτών των δύο διαφορετικών άκρων είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Όταν είναι μια τράπεζα σε κρίση, ο χειρισμός θα είναι τελείως διαφορετικός ε, από ότι όταν έχουμε τραπεζική κρίση. Είναι σημαντικό και όλοι το θέλουμε να προστατεύσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους καταθέτες και τους φορολογούμενους. Αλλά στην πραγματικότητα, σε μια κρίση, δεν μπορείς να τους προστατεύσεις όλους όπως θα θέλες. Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Και πιστεύω ότι η προστασία του, του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα, γιατί είναι προϋπόθεση για να προστατευτούν όσο γίνεται περισσότερο και οι άλλοι δυο, δηλαδή οι καταθέτες και οι φορολογούμενοι. Και αυτό είναι κάτι που θα υποβάλω στην Επιτροπή αυτή είναι επίσης σημαντικό να ανοίξουμε την ευκαιρία για δημόσια παρέμβαση που θα δημιουργεί σταθερότητα όταν έχουμε συστημική κρίση πραγματική. Γιατί αυτό είναι το πρώτο καθήκον, το πρώτιστο. Γιατί το τίμημα, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να δώσει καταστροφικές επιπτώσεις, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ μου φαίνεται ήταν που είπε ότι το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι τον ίδιο το φόβο. Και αυτό νομίζω ότι ισχύει και πρέπει να το συζητήσουμε και όταν μιλάμε για τραπεζική κρίση, γιατί πρέπει να ε, είμαστε σίγουροι ότι θα καταπολεμήσουμε το φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης που είναι το βασικό πρόβλημα σε μια τραπεζική κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα οι ομιλητές μας να μας πούν πώς θα δούμε τις διάφορες κρίσεις διαφορετικού χαρακτήρα και τι είδους μέσα και εργαλεία θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε. Επίσης, να δούμε την χρηματοδότηση εξυγένσης και τα bail-ins. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη εικόνα πώς θα επιλέξουμε το εργαλείο αυτό του bail-in, της διάσωσης με ίδιους πόρους. Το bail-in εργαλείο είναι πολύ καλό, ε, θεωρητικά, γιατί όταν μπει σε πρακτική χρήση δημιουργεί προβλήματα, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Bailin για να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε. Και υπάρχουν διαφορετικές κρίσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά εδώ που πρέπει να τα συζητήσουμε. Τώρα για τη χρηματοδότηση εξυγίανσης. Και εδώ θα ήθελα να μας πείτε τις απόψεις σας σχετικά με το πόσο σημαντικά είναι τα κεφάλαια όταν μιλάμε για τραπεζική κρίση. Αν δούμε την τάξη μεγέθους των κεφαλαίων που χρειάζονται στην πραγματική τραπεζική κρίση, ε, θα αναρωτηθούμε είναι δυνατόν να βρούμε τόσο τέτοια κεφάλαια τόσο μεγάλα. Δηλαδή όταν όλη η οικονομία ε, μιας ε, χώρας θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες. Ε, αν πρόκειται να σχεδιάσουμε χρηματοδότηση κατάλληλη για την εξυγίανση, πρέπει να ξέρουμε πότε θα χρηματο... πώς θα χρηματοδοτήσουμε, πώς και να ξέρουμε και τα όρια, γιατί δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με τα κεφάλαια αυτά εξυγίανσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον στην πρόταση που θα υποβάλω στην Επιτροπή θα πω ότι είναι σημαντικό να έχουμε εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Γιατί αλλιώ σε μια κρίση αν δεν έχουμε εκ των προτέρων χρήματα δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Από την άλλη πώ θα σχεδιάσουμε αυτά τα προγράμματα χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη σήμερα που είναι υπερχρεωμένα. Πώ θα βαθμονομήσουμε τη χρηματοδότηση, πώ θα τη διαβαθμίσουμε σε αυτέ τι οικονομίε. Ε, Αυτά είναι κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση σχετικά με το τι δέον γενέστε καμιά φορά ξεπερνιέται από την ε, αντίληψη ότι αν κάνουμε κάτι λύνουμε το πρόβλημα. Ελπίζω ότι στην ακρόαση αυτή θα ε, παρουσιαστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν και πώς θα κάνουμε το σωστό. Και πάλι χαίρομαι που απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας οι ομιλητές και με ενδιαφέρον θα ακούσω ε, το τι έχουν να μας πούν. Σας ευχαριστώ. Θα στραφώ τώρα στο Πόλο Λούνγκρεν, που είναι Γενικός Διευθυντής του Σουηδικού Εθνικού Γραφείου Χρέους. Α, είστε λίγο μακριά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι πω η πρόσκληση για την οποία σα είμαι γνώμονα οφείλεται στο ότι ω υπουργό διαχειρίστηκα τη δική μα δημοσιονομική και τραπεζική κρίση πριν από 20 χρόνια στη Σουηδία. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ότι είναι κάτι άλλο το να φτιάχνετε τώρα νομοθεσία. Για μένα είναι αναγκαίο να υπάρχει ωστόσο μια συνολική ανάλυση των επιπτώσεων στο τραπεζικό σύστημα και τις εθνικές οικονομίες. Για παράδειγμα, αν δούμε ένα παράδειγμα του εργαλείου Bailin βεβαίω θα αυξήσει αυτό το κόστος του κεφαλαίου και θα επηρεάσει την ανάπτυξη και την οικονομία. Φυσικά υπάρχουν πράγματα λοιπόν που πρέπει να εξεταστούν. Το σημείο εκκίνησης για τη σχόλιά μου και για ε, την πρόταση οδηγία είναι ότι μια κοινωνία χρειάζεται ένα ορθός λειτουργών ε, τραπεζικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κεφαλαϊκή βάση για τις τράπεζες γενικά ω σύστημα. Και, αυτό, και αυτή είναι επαρκή για την πίστοση που χρειάζεται στη χώρα και πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα χρηματοδότηση. Γιατί αν υπάρχει μια βάση κεφαλαϊκή αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, δεν ε, μπορεί να λειτουργήσει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα. Έπειτα μπορούμε να πούμε πως μια συστημική κρίση όπως είχαμε στη Σουηδία πριν από 20 χρόνια θα πρέπει να τη διαχειριστούμε πολύ διαφορετικά από ότι όταν έχουμε ένα μόνο θεσμό που καταραίει. Βέβαια σε σχέση πάντα και με το μέγεθος του εν λόγω οργανισμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συστημικέ κρίσει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο και ορισμένα εργαλεία από αυτά που προβλέπονται από την οδηγία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια συστημική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι χρειάζεται και ευελιξία και αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Αν έχουμε μια συστημική κρίση, είναι αναπόφευκτο ότι οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες κατά συνέπεια θα πρέπει να διαχειριστούν Οι κυβερνήσεις αν υπάρχει συστημική κρίση θα πρέπει να παρέμβουν και να αναλάβουν δράση και πρέπει να αναλάβουν δράση γρήγορα και με διαφάνεια. Αν, είχατε αυτή την κρίση χρέους που αντιμετωπίσαμε εμείς και που αντιμετωπίζουν τώρα οι χώρες της Ευρωζώνης, θα πρέπει να έχεις ένα τραπεζικό σύστημα και μια οικονομία που, όπου θα πρέπει να χειριστεί τα προβλήματα λιτότητας και ανάκαμψης. Και αυτό έχουν πρόβλημα οι κυβερνήσεις να κάνουν, να χειριστούν τις συστημικές κρίσεις. Πρέπει να έχεις περισσότερες εξουσίες παρά εργαλεία που να χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις με τις εξουσίες που έχουν. Βλέπω λοιπόν ότι οι εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην κρίση του 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα δεν υπάρχουν πια σε αυτή την οδηγία. Το ένα είναι οι εγγυήσει για χρηματοδότηση. Δεν μπορείς βέβαια να αποκλείσεις ότι χρειάζεται για να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε ειδική περίπτωση ότι θα χρειαστεί να εγγυηθεί στη χρηματοδότηση, όπως κάποιες φορές χρειάζεται να παρέμβεις και με απόρριψη. Ε, ε, Κι εγώ ήμουν πολιτικός και διατέλεσα για 29 χρόνια πολιτικός και παλιά πίστευα ότι, δεν, ότι μπορούσαμε να χειριστούμε τις τραπεζικές ε, κρίσεις χωρίς πολιτική παρέμβαση, αλλά αυτό δεν ισχύει τελικά. Πρέπει, είναι πολιτικά θέματα αυτά. Πρέπει επίσης να αναλάβει κανείς και να ελέγξει μια ε, καταραίουσα τράπεζα. Με κάποιον τρόπο οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν μια τράπεζα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη μιας της ανάδυσης μιας συστημικής κρίσης και, και να αποφύγουν τον κίνδυνο εξάπλωσης και στις υπόλοιπες τράπεζες. Επίση, θα πρέπει να δει αν υπάρχει δυνατότητα να κάνεις ενέσεις κεφαλαίου και ταυτόχρονα να αναλάβει προσωρινά την, την ε, κατοχή, την ιδιοκτησία. Μπορεί η προσωρινή ιδιοκτησία να είναι για κάποια χρόνια, αλλά σίγουρα όχι για πάντα η διαχείριση, όταν, η διοίκηση μάλλον, όταν χάσει τον έλεγχο της τράπεζάς της, θα καταλαβαίνει ότι πρέπει να συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάσει την τράπεζα. Επίσης θα πρέπει να συμπεριφερθεί με τρόπο ώστε να ανακτήσει και να αποπληρώσει την χρηματοδότηση που έλαβε. Είχαμε 25% ε, χρέος ε, σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά μπορέσαμε με την κρατικοποίηση ή εν πάση περιπτώσει με την προσωρινή κρατική ιδιοκτησία να το αντιμετωπίσουμε. Η κεντρική μας τράπεζα, η κύρια μας τράπεζα λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο ώστε τα, το κομμέριδι και τις... Ε, τα κέρδη μας έδωσαν πίσω όλα τα χρήματα που, μπορέσαμε να, που χρειάστηκε να δώσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολιοξία κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Now, uh, uh, Frank. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Φρανκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναφέρω κάποιες ιδέες μου. Θα περιοριστώ σε τέσσερα σημεία. Ο κύριος Λόμπεν ήδη μίλησε για το μηχανισμό αυτό, για το εργαλείο αυτό που περιέχει μεγάλη ευελιξία. Τα προβλήματα των τραπεζών είναι τόσο διαφορετικά που πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να επιληθούν όλα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και σειρά ρυθμίσεων και κανονισμών. Χαίρομαι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις μια μεταβατική τράπεζα όπως λένε. Τώρα, το αρνητικό αυτής της πρότασης ε, οδηγίας, σχέδιο είναι ότι άσχετα με το αν είναι μεγάλη, μικρή μια τράπεζα, αν είναι συστημική ή όχι, οι κανόνες θα πρέπει να επιβληθούν και να ισχύουν για όλες τις τράπεζες. Πολύ αμφιβάλλω αν αυτό είναι ορθό. Στη Γερμανία έχουμε τον τομέα των ε, αποθεμάτων, τον τομέα των καταθέσεων και τον τομέα των επενδύσεων και πιστεύω ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων γίνεται με πολύ πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι θα το έκανε κατά την άποψή μου μια αρχή κυβερνητική ή κεντρική. Αν λοιπόν μια τράπεζα θεωρείται συστημική, ναι, μπορεί να επέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν όχι όμως, ας αφήσουμε τις περιφερειακές ενώσεις τραπεζών να επιλύσουν τις δυσκολίες. Δεύτερον, το θέμα του bail-in. Bail-in είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε και ξαναχρησιμοποιούμε και εμφανίζεται πολλές φορές σε αυτήν την οδηγία. Την κάλυψη δηλαδή τμήματος του χρέους Πιστεύουμε ότι αν κάποιος προτείνει διαφορετικές μετοχές. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να καλύψει τις ανάγκες ε, και τις επιδημίες πολλών και διαφορετικών ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου τελικά ή του ακάλυπτου χρέους. Αν αυτό το bail τελικά πετύχει, θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην να μην ε, επιδεινώσει τη συστημική κρίση και για τις λεγόμενες ΣΥΦΗ, δηλαδή οικονομικούς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι πολύ μεγάλα για να αποτύχουν, όπως λέμε, too big to fail, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το bail-in ουσιαστικά είναι μια ιστορία διαφορετικής αντιμετώπισης ε, των λογαριασμών. Δεν πρόκειται για νέα χρήματα που ε, ενσωματώνονται σε μια τράπεζα. Είναι όμως ένα σωστό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί αυτό το ακάλυπτο χρέος. Το χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο, το οποίο βεβαίως είναι και πολύ δαπανηρό. Θα πρέπει να αποτρέψουμε τις τράπεζες από την χρησιμοποίηση αυτού του εργαλείου και θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την πρόληψη. Και εγώ θα ενθάρρυνα τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν βεβαίως αυτό το εργαλείο σε περιπτώσεις εκαθαρίσεων ή εξυγίανσης, αλλά θα τους ενθάρρυνα κυρίως να λάβουν μέτρα πολύ πριν, πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ή πολύ πριν ε, φτάσουμε στην ενεργοποίηση ή εντοπίζοντας καλύτερα ποιες είναι οι αιτίες που τελικά παράγουν αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι αυτό το ακάλυπτο χρέος δεν ενσωματώνεται σε άλλες ε, μεγάλες τράπεζες, σύφη, too big to fail, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το απομονώσουμε, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο συστημικό ε, κίνδυνο. Αν γίνει μια άμεση καταστροφή, μια καρδιακή προσβολή παραδείγματος χάνει σε μια τράπεζα, οι άλλες τράπεζες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει η λύση λοιπόν να εξευρεθεί άμεσα, μέσα σε δύο μέρες παραδείγματος χάνει, από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Και ε, μιλώντας με τραπεζίτες διαπιστώνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να προτείνει ένα τέτοιου είδους ε, σχεδίου εξυγίανσης, επανοργάνωσης, αναδιάρθρωσης μέσα σε δύο μέρες όπως θα προβλέπετε σε αυτά τα σχέδια. Σε μια περίπτωση καρδιακής προσβολής, έτσι, άμεσης κρίσης και πολύ ξαφνικής. Γι' αυτό και θα ήταν πολύ πιο λογικό να ενσωματώσουμε κάποια μέτρα προληπτικά και θα πρέπει παραδείγματο χάρη στο κεφάλαιο να ενσωματωθεί πολύ ψηλότερο ποσοστό για την κάλυψη αυτού του χρέους, έτσι ώστε να αποφευθεί το bail Ευχαριστώ, Κρίστιαν Κλάουσεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή τη συνεδρίαση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Τα καθεστώτα εξυγίανσης και διάλυσης είναι κατά την άποψή μου τα πιο σημαντικά ε, στοιχεία στον νέο κανονισμό, ε, ο οποίο είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Είμαι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή ε, Συνομοσπονδία Τραπεζών και μιλώ εξ ονόματο όλων των τραπεζών, μεγάλων, μικρών, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων, τοπικών τραπεζών. Μαζί παρέχουμε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό ακριβώ κοιτάμε να δούμε πώ μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Ε, χρηματοδοτούμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και την κατανάλωση και δίνουμε τη δυνατότητα για απασχόληση και ανάπτυξη. Η στην Ομοσπονδία μας θα υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και αν εφαρμοστεί σωστά θα υπάρξει δυνατότητα ε, ανακεφαλοποίησης μιας τράπεζας ε, χωρίς να δημιουργηθούν συστημικές επιπτώσεις ε, προς άλλες τράπεζες και την οικονομία. Και φυσικά θα διέπουν και τη συμπεριφορά των τραπεζών και θα μειώσουν την ανάγκη να παίρνουμε τα χρήματα των φορολογικουμένων. Ωραία. Αλλά είναι δύσκολο και περίπλοκο. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε απλά τα πράγματα. Όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει ε, ε, κρίση, τα πράγματα συμβαίνουν πολύ γρήγορα. Το γνωρίζουμε πλέον αυτό και επομένω χρειαζόμαστε συγκεκριμένε αρχέ. Μπορούμε να αναλάβουμε δράση και διορθωτικά μέτρα εάν ε, ο κανονισμό είναι αυστηρό αλλά ευέλικτο. Δεν χρειάζονται εκατοντάδε αναλυτικέ οδηγίε για το πώ μπορούμε να προβλέψουμε κάθε περίπτωση. Αν λοιπόν αυτή είναι η φιλοδοξία μας, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για ένα πράγμα. Όταν προκύψει κρίση θα είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε και ένας πολύ αναλυτικός κανονισμός μάλλον θα επιβραδύνει την κατάσταση και δεν θα την επιταχύνει. Κατά την άποψή μου, η οδηγία για τη διαχείριση κρίσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες για να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη διαφορά μεταξύ μιας ε, συστημικής ε, τραπεζικής κρίσης ε, και μιας κρίσης ιδιοσυγκρασίας. Εάν οι τράπεζες επηρεάζονται συνολικά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει εκ των προτέρων αναλυτική λύση. Οι τράπεζες οι οποίες πιέζονται δεν μπορούν να στηρίξουν άλλες τράπεζες και τα μέσα της εξυγίανσης, όπως για παράδειγμα το bail-in, θα είναι επικίνδυνα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε επιπλέον συστημικές επιπτώσεις σε όλο το σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές, ε, διάφανο πλαίσιο ε, για να μπορέσουμε να ε, έχουμε μια λύση και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πάντα το κλειδί είναι η απλότητα. Δεύτερον, στα νέα καθεστώτα το τμήμα της εξυγίανσης είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορέσουμε να έχουμε μηχανισμούς που θα διέπουν τις ε, συμπεριφορές των τραπεζών και επομένω θα πρέπει να είμαστε σαφείς και να υπάρχει κατάλληλη εναρμόνιση. Όταν ε, ε, εξετάζουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία μέσω των νέων κανονισμού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι οι τράπεζες πάντα θα βάζουν και οι ίδιες ε, ε, ε, προστασία στο κεφάλαιό τους πάνω από τα ελάχιστα επίπεδα και επομένω, ε, θα πρέπει η διαχείριση να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να είναι πολύ μακριά από προβλήματα ανάκαμψης και θα πρέπει να μην καταλήξουν σε επίπεδο εξυγίαση. Θα, θα πρέπει λοιπόν ε, να φτάσουν στο επίπεδο της διάλυσης διότι εκεί θα, πρέπει, ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα και δεν θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο και διαχείριση. Άπαξ και υπάρχουν λοιπόν τα κατάλληλα κίνητρα και ε, θα πρέπει η διαχείριση να έχει την εντολή να ε, εξηγειάνει την τράπεζα. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος διάλογος με τις εποπτικές αρχές, αλλά το σκληρό έργο με τη χρήση όλων των μέσων θα πρέπει να γίνεται από τη διαχείριση. Και αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Το τρίτο μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον bail όταν ε, ε, ξεκινάει, παραβιάζεται ε, το κατόφλι από το οποίο ξεκινάει η εξυγίανση, οι αρχές οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τράπεζα θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέσα. Μπορούμε να αντιλήσουμε αρκετά διδάγματα από τα αμερικανικά μοντέλα για το τι συμβαίνει όταν μια τράπεζα θεωρείται ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη. Θα πρέπει να διαγραφεί κεφάλαιο, θα πρέπει να χάσουμε κάποιες ευθύνες και το βασικό ζήτημα είναι ε, το bail-in στην εξυγίαση. Γενικώ οι τράπεζες στηρίζουν αυτή την ιδέα του bail-in. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά ο λόγος είναι απλός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ε, τράπεζες να ε, λύσουν μόνοι τους το πρόβλημά τους. Και επομένως θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν και τους πελάτες τους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν επιπλέον συστημικά σοκ στο χρηματοπιστωτικά συστήματα. Γινόμαστε όλο και πιο ε, σοφοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οικοδομήσουμε το bail Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέσο το οποίο θα μας ε, καθορίζεται σαφώς και έτσι όλοι θα ξέρουν εκ των προτέρων ποια ακριβά ε, μέσα είναι και ποια δεν είναι αν υπάρχουν και άλλες ε, ε, ζημίες οι οποίες επιλέγονται στην κατηγορία του bail-in, μπορούμε να δημιουργήσουμε, ελοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργήσουμε επιπλέον συστημικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ε, μακροπρόθεσμο χρέος, παράγωγα και πολύ μεγάλες καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, στην πραγματικότητα έχουμε μια κύρια ανασφάλιστη χρηματοδότηση που θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα του Μπέιλιν. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυτού του γεγονότος είναι ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα μέσα bail-in θα διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές θα έχουν τιμολογήσει το κατάλληλο επίπεδο κινδύνου και θα έχουν θέσει στην άκρη το κεφάλαιο που απολύτει για να το καλύψουν. Θα πρέπει λοιπόν να μετράμε τη δυνατότητα ε, bail-in ε, σε μια συγκεκριμένη βάση κινδύνου ε, πλήρη και θα πρέπει να έχουμε για παράδειγμα για τις περισσότερες τράπεζες ένα ποσοστό 9 με 10% σε κεφάλαιο και 5 με 10% στο bail-in και γεγονός έτσι, το γεγονός είναι ότι έτσι θα έχουμε ένα πολύ εύρωστο ε, ισοζύγιο. Και έτσι θα μπορούν ε, οι τράπεζες να έχουν ε, βασικό κεφάλαιο το οποίο θα τους επιτρέπει να ε, διαλύσουν οποιαδήποτε τράπεζα η οποία βρίσκεται σε διαδικασία χρεοκοπίας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα κατάσταση των κεφαλαγορών και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη χρηματοδότηση και τις ε, αγορές κεφαλαίων και να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα ε, σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να ε, προσφέρουμε μια λύση. Σε γενικέ γραμμέ στηρίζουμε λοιπόν αυτή τη λύση για την εξυγίανση των τραπεζών, αλλά η πρότασή μα είναι καταρχά να είναι απλό, δεύτερον να έχουμε σαφή και εναρμονισμένα κριτήρια και να επιτρέψουμε σε αυτού που γνωρίζουν καλύτερα τη δουλειά να αποκαταστήσουν μια προβληματική τράπεζα και τρίτον να είμαστε πολύ σαφεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία bail-in. Εάν υπάρχει λοιπόν ένα κανονισμό ο οποίο θα γίνει με το σωστό τρόπο, θα μπορέσουμε μαζί να αποφύγουμε ε, προβλήματα και αυτό ακριβώς ε, σημαίνει να ε, είμαστε ε, προσεκτικοί ως προς την τραπεζική μας εποπτεία. Ευχαριστώ. δεν έχω εγγεγραμμένο στον κατάλογο οι σκιώδεις, και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Ο Φιλίπ. Ο Φιλίπ πρώτος. Thank you. Ευχαριστώ. ερώτηση... Ευχαριστώ. Ερώτηση στον κύριο Κλάουζεν. Πείτε μας λίγο γιατί θεωρείτε τα χωριστά μέσα ή εργαλεία ως επιλέξιμα ή όχι για το χρέος Μπέιλιν. Θέλω να καταλάβω την επιχειρηματολογία σας, το σκεπτικό σας. Ναι, αφού είναι απλή ερώτηση, μου φαίνεται καλό είναι να δοθεί και μια άμεση απάντηση. Όπως είπα, γίναμε πιο σοφοί καθώς δουλεύαμε με το σύστημα αυτό. Είναι σαφές ότι όλα το άλλο παθητικό είναι ε, συστημικό με την ε, α ή β έννοια βραχυπρόθεσμες, δηλαδή δεν θα φύγουν γρήγορα. Οι μεγάλες καταθέσεις είναι συστημικές γιατί τις έχουν οι εταιρείε και δεν θέλουμε οι εταιρείε να χάσουν τις καταθέσεις τους. Τα παράγωγα επίσης ε, μπορούν να είναι συστημικά και αυτά και μας μένει μια κατηγορία που είναι η κύρια χρηματοδότηση. Επίσης είναι σαφές ότι υπάρχει και ε, χωριστή κατηγορία όπως την έχουμε προβλέψει που είναι ευρεία και μετά οι επενδυτές που θα αγοράσουν εκεί ξέρουν τον κίνδυνο οπότε θα βάλουν στην άκρη κεφάλαιο κινδύνου για να την καλύψουν. Μπορεί οι, αυτοί οι ιδιοκτήτες να μην είναι συστημικά σημαντικές, μπορεί να είναι όμως άλλου είδους εταιρείε κεφαλαίου. Θα ξέρουν και θα έχουν βάλει στην άκρη κεφάλαιο κινδύνου και αυτό από μόνο του αποφεύγει, αποτρέπει τους συστημικούς κινδύνους. Η ερώτησή μου έχει εν μέρη απαντηθεί. Γιατί και εγώ ήθελα να ξέρω το εξή. Θέλουμε να προστατεύσουμε το φορολογούμενο, αλλά αν τα ταμεία συντάξεων ε, επενδύσουν σε μέσα bail-in, μπορεί και αυτοί να πάνε γυρεύοντα και στο τέλο να πληρώσουν και αυτοί το λογαριασμό. Πώ θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. στην πραγματικότητα όταν εξαφανιστούν τα κεφάλαια και ε, ε, εδώ μιλάμε για εξυγίανση δεν ε, έχει μείνει τίποτα αφού εξαφανίστηκαν τα κεφάλαια. Τότε θα βάλουμε το μεσο Μπέιλιν διότι θα, πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση θα έχουμε ορίσει ποια θα είναι τα μεσα Μπέιλιν. θα το ξέρουν οι ιδιοκτήτες, αυτοί που θα τα πάρουν, θα επενδύσουν και ε, βέβαια ε, σε, στα ταμεία θέλουν να κάνουν επένδυση με απόδοση των επενδύσεων και μετά θα πρέπει αν τους ενδιαφέρει να δουν ποια είναι, ε, ποιος είναι ο συγκεκριμένος κίνδυνος, πώς τον ε, ετικοποιούν Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε στο τέλος βέβαια θα πρέπει να υποστούν μια απροσδόκητη ζημία. Να πω κάτι κι εγώ γιατί μπαίνει στα δικά μου τα χωράφια που ήθελα να κάνω κι εγώ ερωτήσεις. Έχετε ιδέα για το κόστος αυτών των εργαλείων bail-in γιατί ε, αν υπάρχει ε, η περίπτωση, ο κίνδυνος χρεοκοπίας, τότε θα πρέπει να είναι κοντά στα ίδια κεφάλαια. Έχει γίνει κάποια δουλειά για να ξέρουμε πώς θα εντάξουμε τις, ε, τα προαπαιτούμενα για κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών κλπ. Γιατί ένα πρόβλημα σημερινό που έχουμε είναι ότι υπάρχει διάσωση ή μάλλον απομόχλευση από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων, για να το πω έτσι, λόγω της, ε, των προαπαιτούμενων του Solvency 2. Και αυτά τα μέσα πιστεύετε ότι θα ε, ισχύσουν με τον ίδιο τρόπο και οι ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα μπορούν να επενδύσουν σε αυτά τα καινούργια μέσα και άμεσα συνδεδεμένο με το παραπάνω. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια σύνθετη ιεράρχηση αυτών των μέσων. Εγώ, γιατί είπατε ότι πρέπει να είναι απλό το σύστημα και ότι δεν θέλουμε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αν και έχω δει άρθρα στον τύπο να λένε ήδη ότι υπάρχουν και εφευρίσκονται διαφορετικά επίπεδα αυτών των μέσων. Γιατί ο λιγότερο επαγγελματίας επενδυτής μπορεί να ε, ξαφνιαστεί βλέποντας ότι κρατάει κάτι πολύ επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο από αυτό που νόμιζε ότι έχει. Μπορεί να παγιδευτεί δηλαδή σε ενα μπέιλιν που δεν το ήθελε και δεν το περίμενε. Με απασχολεί αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που προκύπτει σε αυτά τα πλαίσια. Δεν ξέρω αν έχει κανείς μια απάντηση. Να δώσω κάποια σχόλια, να κάνω κάποια σχόλια. Αλήθεια είναι ότι θα υπάρχει κάποιο κόστος εδώ. Ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Τομέας λειτουργεί με κεφάλαια 23. Ε, Όχι, 2-3. Ε, και άλλα δύο θα είναι το κεφάλαιο διάσωσης που θα πρέπει να υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να δούμε αν διατίθεται ως κεφάλαιο κινδύνου. Αν υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια, και αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ τη μια κατηγορία, να ξέρουν αυτοί που επενδύουν ότι δεν θα μπουν σε αυτό τον κίνδυνο. Έχουν γίνει 42 ε, με 80 ε, μονάδες βάσης έξτρα κόστο. Αυτέ είναι οι εκτιμήσει. Είναι ένα σημαντικό έξτρα κόστο. Τώρα, γιατί το κόστο δεν είναι υψηλότερο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μετά την χρεοκοπία θα πρέπει να έχουν κάποιο ε, ε, πριν από το bail-in το κεφάλαιο το συνολικό των τραπεζών θα είναι 12 με 14%. Οπότε ε, αν είναι 12% να ε, γίνει αποσβεστή όταν γίνει εξυγένση. Αυτό έχει ήδη αποσβεστεί και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε όλες τις μεγάλες ε, καταρρεύσει τραπεζών που είδαμε στην κρίση, αυτή ήταν η απώλεια αυτή τη τάξη μεγέθους. Οπότε δεν χάνεται όλο το κεφάλαιο Μπέιλιν, αλλά διατηρείται ω νέο κεφάλαιο για την τράπεζα. Τώρα το, η περιπλοκότητα, το να έχουμε 7 διαφορετικά επίπεδα και κατηγορίες δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε τον Μπέιλιν. Αν βάλουμε εκεί ε, επίπεδα, τότε θα περιπλακεί πολύ η εξυγίανση. Γιατί λοιπόν να μην ορίσουμε ακριβώς τι είναι, ένα μέσον είναι και μετά θα πούμε ότι θα το εντάξουμε σωστά. Γιατί τα δύο, ε, τρεις ε, για το, ε, ως κεφάλαια Μπέιλιν δεν είναι κεφάλαια που μπορούμε να τα βρούμε εν μια ανοιχτή. Τώρα το αν το συνολικό κόστος των κεφαλαίων των, κεφαλαίων, των τραπεζών αυξάνονται ή όχι δεν είναι σαφές όταν κάναμε μια έρευνα για τη μετοχοποίηση σε πολλές δόσεις, είδαμε ότι τα συνολικά δάνεια μειώνονται στη μετοχοποίηση όταν έχουμε πιο διαφοροποιημένα ε, επίπεδα. Υπάρχει λόγος να πούμε λοιπόν ότι και εδώ αν έχουμε πρόσθετες κατηγορίες κεφαλαίων μπορεί στο τέλος να μειωθούν οι συνολικές ε, κεφαλαιακές διαπάνες. Αν δούμε τώρα τα επιτόκια Έχουμε δηλαδή στις τράπεζες ε, διαφορετικά. Είναι υψηλά τα επίσημα επιτόκια, αλλά είναι υψηλά γιατί σε φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει μόνο καθοδική τάση, όχι ανωδική ε, ε στις απαιτήσει. Και αυτό αυξάνει τα επιτόκια. Είναι επικίνδυνο όμως να πάρουμε μόνο τα ε, επιτόκια στην ονομαστική τους αξία. Ένα ζήτημα που δεν το συζητήσαμε είναι σε ποιο βαθμό δεχόμαστε στην ε, οδηγία για τα κεφάλαια μία υποκατάσταση, δηλαδή βασικό κεφάλαιο και bail-in χρέος. Χρειάζεται κάποιο μαξιλαράκι συνολικό, όπως είπε και ο κύριος Κλάουζεν, μια σπίδα προστασίας και υποκατάσταση του συντελεστή για το bail-in στο βασικό κεφάλαιο, στα προαπαιτούμενα βασικού κεφαλαίου, ε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αν ε, ρωτήσω με τις τράπεζες αν είναι ελκυστικό το bail ή όχι. Τώρα, για το ρόλο των συνταξιοδοτικών ταμείων, αρέσκονται πολλέ φορέ να επενδύουν σε ε, επενδύσει ρίσκου. Ε, και βέβαια αυτή η περίπτωση έχει επίσης ρίσκο όπως όμως και πολλά άλλα όπως άλλες κατηγορίες. Δεν είναι το bail-in πιο επικίνδυνο. είναι όπως είναι οι επενδύσεις σε μετοχές. Καταρχήν, όσον αφορά το κόστος, εννοείται ότι μια ισχυρότερη από, από κεφαλαίου τράπεζα σίγουρα θα έχει και καλύτερα πιο ισχυρά εργαλεία για το bail-in και με κόστος χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος θέλει να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο, πρόκειται για μετοχές. Και δεν θα είναι τόσο εύκολο να πει σήμερα κανείς ποιο θα είναι το κόστος αλλά κάποιο κόστος σίγουρα το αναλαμβάνει η κοινωνία. Το θέμα είναι αυτός ο μηχανισμος ε, Μπέιλιν, είναι εύκολο να λειτουργήσει από τη στιγμή που κάποιος γνωρίζει τους κανόνες. Αν πρόκειται για συστημική τράπεζα, παραδείγματο χάρη, ο κύριος Κλάουσε είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες κατηγορίες κεφαλαίου, κάποιοι οργανισμοί που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε μια συστημική κρίση. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το μηχανισμό. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων, ατομικών τραπεζών και συστημικών περιπτώσεων όπου το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο δύσκολα. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Καταρχήν, δεν θέλω να δημιουργήσω αντιπαραθέσεις εδώ, αλλά θα ήταν καλό να σας ακούσουμε και να μας πείτε πού διαφωνείτε μεταξύ σας τουλάχιστον. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον για μας. Θα μας αποσαφηνίσει ίσως κάποια προβλήματα αν δούμε που δεν συμφωνείτε. Όπως είπε ο κύριος Κλάουζερ, τα θέματα αυτά εξυγίανσης, σχέδια εξυγίανσης, εκαθάρισης, θα πρέπει να γίνονται μεμονωμένα, ατομικά ή συνολικά, σε κάποια κατηγορία τραπεζών. Τρίτον, όλοι αναφερθήκατε στο θέμα του Μπέιλιν και των μεγάλων τραπεζών. Όλοι ξέρουν τι είναι συστημικός κίνδυνος. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να το ορίσει. Εκεί γίνεται περίπλοκο το θέμα. Ίσως μπορούμε κάποιος να θεωρήσει ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη τράπεζα. Αλλιώς μπορεί κάποιος να πει ότι πρόκειται για κανόνες που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται σε κάποιες τράπεζες. Αν όμως οι τράπεζες δανείζουν χαμηλότερα ποσά σε τράπεζα, κάποιος άλλος θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτές τις τράπεζες. Και αν οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω του solvency παραδείγματο χάρη δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις τράπεζες, να δανείσουν χρήματα στις τράπεζες, κάποιος άλλος θα πρέπει να το κάνει. Και εδώ ο συστημικός κίνδυνος πάει κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους φορείς και οργανισμούς οι οποίοι καλούνται να δανείσουν. Όταν λοιπόν πλησιάζουμε την κρίση, καταλαβαίνετε ότι η ανησυχία αυξάνεται και το πρόβλημα το 2008 στην κρίση ήταν αυτό, ότι κανείς δεν ήθελε να δανείσει στις τράπεζες και πάγωσε η κίνηση των κεφαλαίων. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό το εργαλείο Μπέιλιν, βεβαίως μου φαίνεται πάρα πολύ αποτελεσματικό έτσι ώστε να είναι έτοιμες να αντιδράσουν οι τράπεζες. Όμως, όμως θα πρέπει να δούμε στην πράξη πραγματικά τι γίνεται. Κύριε Κλάουζε είπατε ότι κάποια κατηγορίες κεφαλαίων πρέπει να εξαιρεθούν. Θα ήθελα να μου πούν οι άλλοι συναδελφοί σας. Ποιες κατηγορίες κεφαλαίου πρέπει να εξαιρεθεί από τον Μπέιλιν. Πριν ε, περάσουμε σε απαντήσεις από αυτού, υπάρχει κάτι άλλο που θέλει να ρωτήσει κάποιος από εσά. Φίλιπ. Ταιριάζει με την ερώτηση του Γκούντερ. Ναι, ήθελα να συνεχίσω σε αυτά που είπε ο κύριος ε, Κλάουσεν. Αν εξαιρέσετε όλα τα άλλα μέσα, δεν ε, πιέζετε τις τράπεζες ε, να αναλάβουν αυτές τη διάθεσή σου και, αφορά το, και να συρρυκνωθούν. Και όσον αφορά το κόστος της κοινωνίας και το τι θα γίνει να το κάνουν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος του να μην ληφθούν μέτρα και την αντιμετώπιση της κρίσης. Και αυτό μάλλον δεν θα βαρύνει τα ίδια άτομα. Θέλετε να μιλήσετε τώρα ή αργότερα. Ίσως καλύτερα να θέσετε την ερώτηση σας τώρα για να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο πάνελ. Ωραία, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Λόγκρεν. Εσείς ήσασταν ένας από τους βασικούς ε, ε, ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλο στη διάσωση της Σουηδίας. Μπορούμε να το πούμε τότε. Εγώ ήμουν στο κοινοβούλιο τότε, ήταν και ο συνάδελφος εκεί, ε, ο Χόκμαρ, δεν τα πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά. Εσείς όμως αναλάβατε δράση και κάνατε κάτι για να μπορέσουμε να σώσουμε την οικονομία. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί διάβασα μία συνέντευξή σας πριν από κάποιες μέρες, Ήσασταν πολύ επικριτικός ε, προς την Τραπεζική Ένωση και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Επειδή είναι μακρά η πείρα θα ήθελα πραγματικά να ακούσω γιατί είστε τόσο επικριτικός και τι εναλλακτική λύση θα προσφέρατε εσείς. Ωραία. Εάν ε, μπορείτε να απαντήσετε. Δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο πρώτος. Ο κύριος Λάγκρεν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ απλή ερώτηση. Ποια είναι η εναλλακτική λύση στην Τραπεζική Ένωση. Νομίζω και ελπίζω εν ευθέτω χρόνο να υπάρχει μια ε, κοινή προσέγγιση, ε, δηλαδή να υπάρχουν και άλλες ενώσεις ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ εντάχθηκα στο κόμμα μου γιατί είμαι υπέρ της Ευρώπης. Θεωρώ όμω ότι αυτοί που χαράσουν πολιτική στην Ευρώπη να συζητήσουν ποια είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε λύσεις για να σώσουμε τις ε, ισπανικές τράπεζες και ταυτόχρονα να γίνει μια διαρθρωτική συζήτηση για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέε δομέ στο ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την άποψή μου δεν ε, λύνει τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λύσουμε ε, αυτά τα οποία μας απασχολούν περισσότερο. Δεν διαφωνήσαμε και πάρα πολύ νομίζω με το συνάδελφο, απλώ έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. μπορεί να ενισχύσουμε τις τράπεζες, αλλά κατά την άποψή μου μπορεί να υπάρχει και πρακτικό κόστος για την κοινωνία και θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα ε, αναλυφθεί αυτό το κόστος. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μελέτες. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφωνία μας. Αυτό όμως το οποίο συμφωνούμε είναι το πιο ενδιαφέρον. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει απλή νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε ε, διάφανη, να είναι σαφή τα πράγματα και να υπάρχει και αυτή η ελαστικότητα που επιτρέπει στις κυβερνήσεις όταν προκύψουν συστημικές κρίσεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, το too big to fail δεν σημαίνει ότι αναφερόμαστε μόνο στις μεγάλες τράπεζες. Ε, είχαμε προβλήματα και με τις μικρές επενδυτικές τράπεζες στη Σουηδία το 2008, γιατί μετά τη Lehman Brothers υπήρχαν προβλήματα και για αυτές τις μικρές τράπεζες. Μπορεί να δημιουργηθεί κρίση λόγω αύξηση των επιτοκίων και το καθεξής. Εξαρτάται λοιπόν και από το όλο, ε, την όλη περιραίωση ατμόσφαιρα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ μία συγκεκριμένη ερώτηση σε επίπεδο καθάρισης, σε επίπεδο μήλων. Ε, είναι λογικό να γίνεται σε επίπεδο μήλων. Αμφιβάλλω κατά πόσον μπορεί να γίνει σε επίπεδο νομικών προσώπων, ιδίω ε, για τράπεζε ε, που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά σε διάφορε χώρε. Και αυτή είναι και η συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα με τον κύριο Ένερια. Το να υπάρχει ένα σώμα εποπτικό είναι πολύ σημαντικό να αποφασίζει συλλογικά αυτό το σώμα γιατί πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και οι χώρες πρέπει να δέχονται τις αποφάσεις ε, που ε, λαμβάνονται από το σώμα σε επίπεδο ομίλου για να σωθεί η τράπεζα. Για τις παγκόσμιες ε, συστημικές τράπεζες ετοιμάζουμε θέματα εκαθάρισης και εξυγίανσης και είναι σημαντικό το ποσό στην εξηγήση και αντίστοιχο ποσό θα έχουμε και στην εκαθάριση. Και το να γίνει αυτό για ελάχιστες χώρες ε, δεν είναι δυνατόν και θα υπάρξει πρόβλημα ε, για τις ε, χώρες που θα χρειαστούν να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα σε, σε συλλογικό επίπεδο. Ακόμα και ένα ενιαίο επόπτη ε, θα μπορούσε να αποφασίσει σε συλλογικό επίπεδο, που συζητήσαμε νωρίτερα σήμερα. Καταρχάς, οι τράπεζες Οι τράπεζες δεν θα κάνουν ποτέ βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και πριν από την κρίση. Ε, δεν ε, λύνει το πρόβλημά μας και δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό. λέτε κατά πόσον υπάρχουν άλλες συστημικές ζημίες. Κάποιες ε, ε, όταν οι τράπεζες δεν έχουν τα χρήματα ε, μπορεί να μην είναι, αλλά οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να χαθούν καταθέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν θα πρέπει ξαφνικά να πάνε στο κεφάλαιο της τράπεζας. Αυτό θα είναι συστημικός κίνδυνος. Όσον αφορά το θέμα των συστημικών κινδύνων, είναι πολύ δύσκολο να το καθαρίσουμε, αλλά αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι όταν δεν αναγνωρίζεται ο κίνδυνος ή όταν δεν καθορίζεται ότι αυτό είναι κίνδυνος και δεν ε, τίθεται ε, στο αποθεματικό κεφάλαιο, τότε δεν μπορούν να ε, απορροφηθούν σε συνέχεια τα κεφάλαια. Εάν όμω καθορίσουμε ποιο είναι ο κίνδυνο και υπάρχει κεφάλαιο στην άκρη, τότε αν υπάρξει απώλεια, τότε μπορεί να γίνει εισρωή κεφαλαίου και δεν έχουμε και μεταφορά και σε άλλου τομεί. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, ε, να καθορίσουμε σαφώς ποιοι είναι οι κίνδυνοι και να υπάρχουν και σχετικά κεφάλαια. Όσον αφορά τα σχέδια εξυγένσης, εκαθάρισης και αν θα λειτουργήσουν ή όχι, αν θα είναι αποτελεσματικά. Εγώ θυμάμαι ότι η Fed, η Κεντρική Τράπεζα στις ΗΠΑ, ήταν πολύ απογοητευμένη όταν είδε πώς αντέδρασαν οι τράπεζες στις Ηνωμένε Πολιτείε χωρίς να μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα. Το θέμα είναι να έχουμε τις πληροφορίες, να λάβουμε τα μέτρα αυτά και να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι. Τώρα ποιος θα χρηματοδοτήσει τις τράπεζες. Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που μάθαμε μετά το 2001 είναι ότι η πραγματική οικονομία δεν υπέστη πλήγματα. Τελικά είδαμε ότι τα νοικοκυριά είναι αυτά που υπέστησαν το πλήγμα και το βάρος και όχι οι τράπεζες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή η μετατροπή σε μετοχές από τις τράπεζες ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε και αυτό ήταν το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο επίπεδο κεφαλαίου όπου σε περιπτώσεις τέτοιων κρίσεων στο τραπεζικό σύστημα τελικά να μην πληρώνουν μόνο τα νοικοκυριά, αλλά ενδεχομένως ή μεσάζοντες όπως ε, τα διάφορα ταμεία. Θα πρέπει δηλαδή να απομονωθούν από τη μία οι τράπεζες και οι ε, ασφαλιστικές εταιρείες έτσι ώστε να εξαιρεθούν κάποιες κατηγορίες από αυτές ε, τις απώλειες. Βεβαίως υπάρχουν και οι διαιτητικές αρχές που παίρνουν κάποιες αποφάσεις ποιος θα προστατεύεται και ποιος όχι. Ναι, αυτό είναι μια επιλογή που πρέπει να γίνει. Και βεβαίω όλε οι τράπεζε θέλουν να μπουν σε αυτή την κατηγορία των προστατευμένων. Ακόμα λοιπόν και αν αποκλείσουμε αυτό το βραχυπρόθεσμο ε, χρέος, θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό το κάνουμε αυτό, 100%. Γιατί κάποια χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμη χρειάζεται με έναν ποσοστό 15-20% έτσι ώστε το κόστος να είναι τόσο υψηλό που να αποθαρρύνουμε αυτή την βραχυπρόθεσμη δανειοδοτική δραστηριότητα. Άκουσα επίσης κάτι που είπατε στην αρχή. Από τη μια χρειαζόμαστε αυτή την εξυγίανση, αυτή την εκαθάριση. Γιατί πόσο όμως μιλάμε, 200-300 δις Πιστεύω ότι πρέπει να είναι τόσο υψηλό το ποσό που να μπορεί να καλύψει πιθανό ακάλυπτο χρέος και απώλειες. Ο φορολογούμενος δέχεται να αναλάβει αυτό το ρίσκο το τραπεζικό σύστημα και τελικά να υποφεληθεί η κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει ο φορολογούμενος ναι μεν να παίξει εδώ κάποιο ρόλο εγγύτη, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό ποσό 80-100 δις και επιπλέον να αναλάβει και κάποιο ρίσκο και ο φορολογούμενος. Θα ήθελα να πω στον κύριο Φράγκη, ότι μιλήσατε για το 2001 την κρίση τότε και την φούσκα. Τότε, βεβαίως, το θέμα του δανεισμού δεν λύθηκε. Τότε είδαμε ότι τα νοικοκυριά ήταν αυτά που αντιμετώπισαν αυτές τις ε, κρίσεις και είδαμε ότι από το 99 παραδείγματος χάρη στη Σουηδία οδήγησε σε μια πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης και γι' αυτό και τα <laughs> μέτρα λιτότητας βεβαίως δεν το λέτε εσείς, αυτό το λέω εγώ, δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόεδρος, τι άλλο θέλετε να ακούσετε από τους εμπειρογνώμονες. Εγώ προσπάθησα να τους προκαλέσω Ίσως ήμουν υπερβολικά ευγενικό όταν ρώτησα αν ε, συμφωνούν ή διαφωνούν μεταξύ τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το μέσο το έχουμε συζητήσει αρκετά, αλλά θα είναι ενδιαφέρον τελικά να ακούσουμε τι έχουν να πούν, καθώς συζητάμε την ευκαιρία για προσωρινή, τη δυνατότητα για προσωρινή ε, κρατικοποίηση και πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει, πώς μπορεί να μπει στην νομοθεσία κάτι τέτοιο. Ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Είπα στην ομιλία μου ότι Όταν είμαστε σε σημείο μη βιωσιμότητα και άρα σε, μπαίνει σε καθάρεση, τότε θα πρέπει ε, η αρχή καθάρισης να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη θέση Ένα παλιό ε, μέσο που υπάρχει, όπω ανέφερε ο Πολ στη Σουηδία, η Σουηδία το έκανε σε αρκετέ περιπτώσει. και πρέπει να πάρει την ε, ιδιοκτησία, να κρατικοποιήσει, να αποφασίσει πως είναι το καλύτερο μέσο ή διαφορετικά χρηματοδότηση ή κεφάλαιο. Γιατί ε, όταν γίνεται καθάριση πάει η τράπεζα. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ε, πάνε, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης, οπότε κάποιος νέος θα, θα έρθει. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να ε, πτωχεύσει και να μην μπορεί να παρέχει πια τις υπηρεσίες της στην κοινωνία η τράπεζα αυτή. Γι' αυτό και πιστεύω πως αυτή η φάση η καθάριση είναι σημαντική, γιατί με τα δάγματα που έχουμε αποκαμίσει και με τις απαιτήσεις της CRD4 οι τράπεζες θα ε, κρατήσουν τη γραμμή όχι μόνο για την καθάριση αλλά και για το σημείο ανάκτησης. Θα υπάρχουν περισσότεροι φραγμοί ώστε να αντιμετωπιστεί νωρίτερα ο κίνδυνος. Και γι' αυτό θα πρέπει και οι αρχές να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία που, που γίνεται. Ναι, και εγώ Συμφωνώ. And Αν ε, ε, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση καθάρισης, ε, χρειάζονται και μετρητά. Το bail δεν μπορεί να δώσει χρήματα μετρητά. Ποιος δίνει μετρητά, η κυβέρνηση ή κάποια τράπεζα κρατική. Πάντως δεν γίνεται να βγει κανείς από την προσωρινή κρατικοποίηση, τη ρητή ή την άρρητη. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά με διάφορους τρόπους, αλλά... Ε, χρειάζεται η δυνατότητα προσωρινής κρατικοποίησης. Μπορούμε να κάνουμε ένα είδος ρήτρα ε, ε, ώστε εάν το σύστημα λειτουργήσει καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε, ο φορολογούμενος μπορεί να πάρει κάποια λεφτά πίσω. Στη Γερμανία το προσπαθήσαμε. Το προσπαθήσαμε με το πρόβλημα των ε, κακών τραπεζών και των ε, επενδύσεων σε ακίνητα. Εάν η κακή τράπεζα λοιπόν την αναλάβει μια καλή τράπεζα, αυτή εξηγιανθεί και εντωμεταξύ μπορεί να επιστραφεί πάλι στην, ε, στην αρχική της κατάσταση μετά από μια μεταβατική περίοδο. οι μεταβατικές τράπεζες όντως μπορούν να είναι ε, μία λύση γι' αυτό και είπα, ε, το χρησιμοποίησαν. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι οι κυβερνήσει να καταλάβουν ότι εφόσον έχει να αντιμετωπίσει μια συστημική κρίση, ε, λείπει η εμπιστοσύνη και όλο ένα και μειώνεται η εμπιστοσύνη. Και αυτό επηρεάζει το ισοζύγιο τη τράπεζα, η οποία είναι πολύ πιο διστακτική στο να δανείσει στον κόσμο που το χρειάζεται. Πρέπει λοιπόν να παρέμβει και να πει ε, ότι πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του ισοζυγίου για να δούμε αν υπάρχουν ανισορροπίες κεφαλαίων για να αποφύγουμε την πάυση των πιστώσεων. Δηλαδή θα πρέπει να εκτιμηθούν τα, κυβερνητικά, τα κρατικά ομόλογα στο σωστή τους αξία και όχι 100% πάνω. Να πούμε λοιπόν, καλύψτε αυτή την τρύπα, να, να επανισορροπηθεί η, το έλλειμμα. Διαφορετικά πρέπει να παρέμβουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν κάθε φορά ποια είναι η κατάσταση και να ζητήσουμε κεφάλαια. Εάν δεν παρέμβουν οι ιδιώτες θα πρέπει να παρέμβουν οι κυβερνήσεις δεχόμενες και την ευθύνη για την κρατικοποίηση, ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να πάρουν και τα χρήματά τους πίσω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να έχουμε και ένα χρόνο για ερωταπαντήσεις. Αν έχετε κάποιες περαιτέρω σκέψεις που θέλετε να μας στείλετε, με τα χαρά θα τις λάβουμε και θα τις διανύμουμε και στους ε, ε, συναδέλφους. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο μας πάνελ που έχει να κάνει με την καθάριση, τη χρηματοδότηση και την, την ε, ε, ευθύνη των εταιριών. Και έχουμε διάφορους εκπροσώπους. Ο Ντάνιελ Γκρός από το ΣΕΠΣΕ και ο Μάριο Νάβα. Ποιος θα λάβει το λόγο πρώτος. Ο κύριος Γκρός. Ήλπιζα ο Μάριο να μιλήσει πρώτος για να του κάνω κριτική αλλά δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται. Μου αφαιρέσατε τη δυνατότητα. Είμαι λίγο μπερδεμένο μετά από αυτή τη συζήτηση που προηγήθηκε με τους ομιλητές, ιδιαίτερα ακούγοντας τη λέξη συστημικός. Συστημικός τι θα πει. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει σε εθνικό επίπεδο, αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει κάτι διαφορετικό σε ενωσιακό επίπεδο. Οπότε όταν μιλάμε για εξυγίανση, νομίζω ότι το θέμα κλειδί είναι ποιο πλαίσιο έχουμε κατά νουν. Ένα που στηρίζεται στην εθνική ανάληψη ευθύνης ή ένα άλλο που στηρίζεται στην Ευρωζώνη και στην μεγάλη της αγορά και σε αυτό που πάμε να ε, κάνουμε την Τραπεζική Ένωση. Γιατί πολλές τράπεζες ή ε, πολλοί τραπεζικοί όμιλοι που θα ήταν συστημικοί σε επίπεδο εθνικό φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πια συστημική αν κρυθούν σε ενωσιακό επίπεδο. Ε, στην Ισπανία ε, οι κάχαση είναι συστημικές για το εθνικό επίπεδο γιατί το δημοσιονομικό βάρος είναι υπερβολικό, δυνητικά τουλάχιστον, ενώ αν λειτουργούσαν σε επίπεδο ένωσης θα ήταν μεγάλο πλήγμα, όχι όμως θεωρούμε συστημικό στην Ευρωζώνη. Θα έλεγα λοιπόν ότι όσο ψηλότερο το επίπεδο που λειτουργεί η αγορά και η χρηματοδότηση και η αρχή για την εξυγίανση, τόσο περισσότερο διαφοροποιείται ο κίνδυνος και τόσο πιο πολύ θα μπορούμε να εφαρμόζουμε καθεστώτα εξυγίανσης και να βάζουμε τους πιστωτές ε, στο Μπέιλιν Σε εθνικό επίπεδο έχουμε θεωρητικά καλά προσδιορισμένοι, θεωρητικά τουλάχιστον, ε, νομικές απαιτήσεις, αλλά de facto ε, υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο ο καθορισμός και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες μέλη είδαμε όπως είπε κάποιος ότι αν τα μέσα τα, κρατα... τα κρατούν συνταξιδοτικά ταμεία ή άλλοι τότε η κυβέρνηση λέει εδώ έχουμε δηλαδή αριστερή τσέπη, δεξιά τσέπη. Ή θα τα δώσω στην τράπεζα για να τα δώσει με τη σειρά τη στα συνταξιοδοτικά, ή δεν τα δίνω στην τράπεζα και θα κάνω μετά διάσωση του συνταξιοδοτικού ταμείου. Αν ο στόχο είναι να εξοικονομήσουμε χρήματα για το δημόσιο τομέα, τότε νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ποιο κρατάει στα χέρια του αυτά τα μεσα μπέιλιν, όπω λέγαμε και πριν. Και πάλι, αν είναι σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου το, τα μέσα bail-in που ε, εκδίδονται από εθνικές τράπεζες θα διακρατούνται ως επιτοπλίστων από εθνικά ιδρύματα, είτε είναι νοικοκυριά, είτε συνδεξιδωτικά ταμεία, είτε οτιδήποτε, κυρίως γιατί είναι πιο κοντά και γνωρίζουν το ρίσκο καλύτερα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ενώ αν έχουμε πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση και αν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που διακρατούν τα μέσα είναι πολύ διαφοροποιημένοι, οπότε να, ένα συνταξιδοτικό ταμείο να έχει ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο όταν υπάρξει πρόβλημα τότε θα πληγούν, αλλά ο κίνδυνος θα κατανεμηθεί σε πολύ ευρύτερο τομέα. Και αυτό είναι ένα όφελος από τη διαφοροποίηση και ε, κατάτιμηση του κινδύνου. Θα έλεγα λοιπόν ότι στο βαθμό που κρατάμε τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και την εθνική χρηματοδότηση για αυτά, άμα τα κρατήσουμε, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες κρίσεις που θα είναι de facto συστημικές και μπορεί να ξαναυπάρξει η αρνητική ανάδραση που είδαμε σε πολλές χώρες. Να είναι σαφές ότι όποτε έχουμε συστημική τραπεζική κρίση, συνήθως η οικονομία πάει πολύ άσχημα και συνήθως και το κράτος αντιμετωπίζει δυσκολίες γιατί αν το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί τότε και το κράτος δεν μπορεί να εισπράξει τους φόρους που πρέπει και κατά πάσα πιθανότητα και το ίδιο θα αντιμετωπίσει δυσκολία. Και θα έχουμε τεράστια εθνικά ταμεία εξυγίανσης τα οποία απαιτούνται για επενδύσεις στο εξωτερικό όμως ούτως ώστε να έχουν κάποια χρησιμότητα ε, σε τυχόν μεγαλύτερη κρίση. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό το βασικό θέμα και λέω, εάν σχεδιάζεται με αρχές και αρμοδιότητες εξυγίανσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι έξω από μικρά ιδρύματα. Το 90% ε, εξαρτάται από το αν κοιτάζομαι το εθνικό επίπεδο ή το επίπεδο ευρωζώνης. Η δυνατότητα αντιμετώπισης της κρίσης και της ανάσχεσής τους για να μην γίνουν συστημικές ε, είναι μεγαλύτερε στην Ευρωζώνη από ό,τι στο εθνικό επίπεδο και μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί στα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τα συστήματα και μέσα bail-in από ό,τι θα είμαστε στο εθνικό επίπεδο. Όποιες και αν είναι οι, όποιοι και αν είναι οι κανονισμοί που ισχύουν στο εθνικό επίπεδο. Σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε στη συνέχεια. Ο κύριος ε, Νάβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλου, και σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τρία είναι αυτά τα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχά, η γενική εικόνα, το σύστημα εκαθάριση αναφέρθηκαν όλοι σε αυτό και χαίρομαι που ο κύριο Όκμαρ και ο κύριο Κλάουσεν είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των όσων προσπαθούμε να κάνουμε. Συμφωνώ απολύτω. αλλά αυτό το σύστημα δεν θα πρέπει να το δούμε μεμονωμένα. Θα πρέπει να δούμε αυτή την πρόταση την οποία κάναμε λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα άλλα στοιχεία που έχετε ενώπιόν σας ε, και συζητούνται σήμερα, διότι οι σχέσεις είναι σημαντικές και οι αλληλεπιδράσεις, όχι μόνο σε υψηλό επίπεδο, αλλά και όταν ε, πάμε να καταρτήσουμε τις λεπτομέρειες. Και αυτό ισχύει και για το CRD και για την ε, Τραπεζική Ένωση και μπορεί να ισχύει και για την ε, συνέχεια, εάν και εφόσον υπάρξει συνέχεια για το θέμα αυτά, διότι τα θέματα τα οποία έθιξε ο συνάδελφος τα έχει θίξει και η ομάδα Λικάνεν. Ε, όλα τα προγράμματα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας, ε, τα ταμεία διάσωσης ε, και τα θέματα της εκαθάρισης είναι αυτά τα οποία μας αφορούν περισσότερο. Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις σύντομες πτυχές. Καταρχάς, τη σημασία των εναρμονισμένων κανόνων για όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι, όπως ακούστηκε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα αμάλογαμα πιθανών εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να είναι εναρμονισμένοι οι κανόνες, διότι αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει να αποφύγουμε ε, κατακαιρματισμό της ε, εσωτερικής αγοράς ε, και μεμονωμένους συμμάχους και να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ κρατών και τραπεζών. Και επίσης ε, θα ήθελα να συνεχίσω και σε αυτά που είπε ο εισηγητής ε, Όκμαρ. Ε, είτε έχουμε εκ των προτέρων χρηματοδότηση, είτε ελοχεύει ο κίνδυνο να μην έχουμε καμία χρηματοδότηση. Εδώ υπάρχει αυτό το θέμα του 1% το οποίο έχουμε προτείνει. Θα ήθελα να το θίξω νομίζω ότι προκειμένου να κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση για αυτό το 1% θα πρέπει να δείτε αυτό που σας είπα στην πρώτη μου παρατήρηση. Αυτό το 1% δεν είναι μεμονωμένο, υπάρχουν και άλλα μέσα τα οποία είτε μειώνουν την πιθανότητα να πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτά τα μέσα, είτε μειώνουν τις επιπτώσεις. Ε, δηλαδή, όταν κάποιος ε, πρέπει να ανατρέξει σε αυτά τα μέσα, θα πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία στο μεταξύ. Και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το bail-in, το οποίο περιλαμβάνεται στην οδηγία μας και με χαρά άκουσα σήμερα το πρωί θα την απεκαλέσω μια συνολική αποδοχή των βασικών αρχών με βασικά δύο ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε και ίσως αυτή η συζήτηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία. Το ένα ερώτημα είναι αν θέλουμε να έχουμε στοχευμένη ή μια ευρύτερη διαδικασία bail-in και αυτό ε, προκύπτει και από την έκθεση Λικάνεν και εκεί υπήρχε ένα πολύ καλό επιχείρημα. Είναι ένα θέμα προ... για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν έχει επιλήξει την ευρύτερη διαδικασία αλλά με χαρά μπορούμε να εξετάσουμε και τα αντίθετα επιχειρήματα και επίσης υπάρχει και το άλλο σκεπτικό ότι ενώ μεν δεχόμαστε τη γενική ε, αρχή θα έπρεπε ίσως να εξαιρέσουμε κάποιες κατηγορίες, ε, ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λύσεις. Μου, άρεσαν οι παρατηρήσεις του κυρίου Φράνκε, ότι θα πρέπει να θυμηθούμε τι είναι αυτό το bail-in. Ε, μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις ένα μερίδιο και επομένως ε, καλό θα ήταν μια μετοχή. Επομένως καλό θα ήταν να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. άκουσα και κάτι αρκετές φορές και από τον κύριο Όκμαρ και από όλους εδώ στην αίθουσα σήμερα το πρωί το θέμα της ε, προσωρινής δημόσιας ιδιοκτησίας. Εδώ νομίζω ότι το θέμα της κράτησης είναι πολύ σαφές. Όλοι όσοι μίλησαν ε, ε, είδαν ποιο είναι το, το αντάλλαγμα. Ανταλλάσσουμε το ιδανικό, αυτό το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε και την πραγματικότητα, αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η η ανταλλαγή και θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε ε, να επιτύχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι είτε δεν θα κάνουμε κάτι που θα κάνει την πραγματικότητα απίθανη ή θα συμβαίνει συνεχώς το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε πού θα βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και κάτι το οποίο γνωρίζομαι ότι θα αποτελέσει θέμα συζήτηση, Είναι το θέμα του αμοιβαίου δανεισμού. Είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στην πρότασή μας. Ακούσαμε ε, αρκετά σχόλια για το θέμα αυτό και θα ήθελα να το συμπεριλάβουμε και αυτό στη συζήτηση. Εν κατακλείδη, ναι, εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα νομοθετήματα τα οποία θα ε, αλλάξει την πορεία της Ευρώπης και μάλιστα για τα καλά. Μπορεί, ελπίζω κάποιος σε 20 χρόνια να έρθει εδώ και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε πριν από 20 χρόνια είχαμε κρίση στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν κάποιος βρίσκεται εδώ μετά από 20 χρόνια και μιλάει για αυτό το πράγμα θα είναι και γιατί ε, το συγκεκριμένο ε, νομοθέτημα μας βοηθάει αλλά όχι μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε και τα υπόλοιπα και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι θα πρέπει να ε, εγκρίνουμε αυτή τη δέσμη μέτρων πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτηση, ο Φιλίπ. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που είπε ο Ντανιέλ Γκρός, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά θέλουμε ένα σχήμα που να καλύπτει όλη την Ευρωζώνη και ιδιαίτερα για τις ε, συστημικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι κάπου, κάπου υπάρχει ένα σύστημα που θα λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει στο τέλος ένας μηχανισμός. Εσείς μιλήσατε για τον Ευρωπαϊκό Σταθροποιητικό Μηχανισμό. Αν όμως υπάρχει υποχρέωση για ομοφωνία στην ψηφοφορία, αυτό σε μια περίοδο κρίσης μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο, μειονέκτημα. Το θέμα της πολιτικής ένωσης βεβαίως, που φυσικά δεν συμπεριλαμβάνει μόνο αυτό το τομέα αλλά και πολλούς άλλους, και μιλήσαμε και για το δημοκρατικό έλεγχο, τη λογοδοσία. Εδώ ουσιαστικά αναλαμβάνουμε για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους ένα σαφές ε, δημοσιονομικό ρίσκο. Είπατε κάτι που με ξάφνιασε. Κατάλαβα ότι αυτό που πήγατε να πείτε είναι ότι για το Λίκανεν για την έκθεση αυτή θα, υπάρξει, θα υπάρξουν και ε, νομοθετικές συνέπειες. Συμφωνείτε, κατάλαβα καλά γι' αυτό, ναι ή όχι. Τώρα, όσον αφορά αυτή την εξυγίανση, διάσωση, τα συστήματα πληρωμών θα πρέπει εδώ να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να τα απομονώσουμε από τις τράπεζες σαν μόνιμη λύση, έτσι ώστε να αποφύγουμε μία τραπεζική κρίση να οδηγήσει σε κατάρρευση κάποιων βασικών υπηρεσιών. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε σε άλλες. Να απαντήσω στον Φιλίπ Λαμπέρα. Κοιτάξτε εδώ είδαμε τους ευρωτεχνοκράτες να φοβούνται ως συνήθως και βεβαίως υπάρχει η αρχή της συλλογικότητας στην Επιτροπή και της απόφασης ε, με συλλογικό τρόπο. Η έκθεση Λίκανεν, ναι βεβαίως ε, πρέπει να σας πω ότι υποστηρίχθηκε και από τον Επίτροπο και από τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Τώρα, αυτή η ιδέα που θέσατε, βεβαίως και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείτε, η έκθεση Λίκανεν για άλλη μια φορά την αναφέρει αυτή την πρόταση σε μια μικρή παράγραφο κάπου στην έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη έχουμε στην Ευρώπη έχουμε διαχωρισμό εδώ των συστημάτων πληρωμών, κάτι που έχει συζητηθεί πολλές φορές σαν ιδέα. Υπάρχει οδηγία όσον αφορά το settlement finality, όπως ήταν ο τίτλος της οδηγίας αυτής, και το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί, αν είναι αρκετή η ασφάλεια που παρέχει ή αν πραγματικά χρειάζεται σαφής διαχωρισμός. Πιστεύω ότι σε κάποια σχέδια μελλοντικά εξυγίανσης, διάσωσης, εκαθάρισης θα πρέπει ίσως να ξανασκεφτούμε αυτό το σαφή διαχωρισμό. Τώρα, ποιος θα είναι ο δημοκρατικός ε, ε, ε, ε, η δημοκρατική στήριξη. Και όσο ο Ευρωπαϊκός Σταθεροποιητικός Μηχανισμός λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να υπάρξει και να λειτουργήσει η δημοκρατική στήριξη. Το θέμα είναι να δούμε αν εδώ η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από κοινού. Προς το παρόν όμως παραμένει εθνική χρηματοδότηση. Μέχρι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μεγάλο ταμείο για τις πληρωμές, για το σύστημα πληρωμών, θα συμφωνήσω με τον Μάριο. Ε, Θα συμφωνήσω με τον Μάριο έλεγα για τις πληρωμές αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ειδωθεί αυτό τελείως ξεχωριστά και την μπαίνουμε σε πάρα πολύ, πάρα πολύ ε, δύσκολες ερωτήσεις και πρόεδρος ο Φιλίπ έκανε και μια ερώτηση στους προηγούμενους ομιλητές με εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν εφαρμόζουμε εδώ την αρχή της επικουρικότητας, όπως είπε και κάποιος άλλος ομιλητής. Εδώ έχουμε δίκτυα ασφαλείας σε κάποιες χώρες για το τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτές τις τραπεζικές τις ενός τραπεζών να διευρύνουν το φάσμα αυτών των δικτύων ασφαλείας έτσι ώστε κάποια προβλήματα να ενσωματωθούν σε αυτά. Πώς μπορούμε όμως, και εδώ είναι το ερώτημα, να απομονώσουμε τις τράπεζες από τις εθνικές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα που προϋποθέτει πολύ στενή συνεργασία και σχέση μεταξύ τραπεζών και κυβερνήσεων. Εγώ λοιπόν εδώ θα ζητούσα περισσότερα δίκτυα ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα. Δεν αρκεί εδώ ούτε ο περιφερειακός ούτε ο εθνικός ε, τομέας και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει το υπόλοιπο πρόβλημα να καλύπτεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος, ποιος άλλος ήθελε να πάρει το λόγο. Ένα σχόλιο όσον αφορά αυτό το διαχωρισμό. Για μένα είναι σαφές ότι η Ευρώπη έχει μεγάλες τράπεζες οι οποίες έδειξαν ότι έχουν το μέγεθος να επιβιώσουν από αυτή την κρίση. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί για αυτές τις περιπτώσεις όπως και ο κύριος Νάβα θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε σε αυτές τις τράπεζες το λεγόμενο implicit capital, κέρδος κεφαλαίου. Και εδώ θα πρέπει να δούμε κάτι που μέσω των νέων τεχνολογιών αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, το, τις πληρωμές, οι οποίες είναι ένα συνολικό σύστημα ηλεκτρονικών, αν θέλετε, διευθετήσεων πληρωμών. Οι συναλλαγές γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, όλες οι εγγύσεις. Όλα λοιπόν είναι αλληλένδετα. Και δεν μπορούμε εδώ να λειτουργήσουμε με ιδέες και τεχνικές του παρελθόντος χρόνου. Σήμερα χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα για να γίνουν οι πληρωμές. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει εδώ να εγγυηθούμε και να διασφαλίσουμε είναι ότι εγγυόμαστε τη λειτουργία μιας τράπεζας. Και γι' αυτό και μιλάμε για εξυγίανση σε περίπτωση δυσκολιών, εκαθάριση κτλ. Και αν υπάρξει απώλεια κεφαλαίου, κάποιες διευθετήσεις. Πρόεδρος, η Ελίζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις ε, του πάνελ για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Δεν έχω αμφιβολίε για το πώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμό σε φυσιολογικού καιρού, όχι σε εκτακτή ανάγκη. Με, με την ομοφωνία για την αντιμετώπιση μεμονωμένων τραπεζών και κατά πόσο θα έπρεπε να είναι ένα μέσο για τη φάση καθάρισης ή ανακεφαλαιοποίησης. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Για στο ίδιο θέμα ο μηχανισμός σταθερότητας θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα στήριγμα για τα κονδύλια ε, τα εθνικά κονδύλια καθάρισης για τις μεμονωμένες τράπεζες να αποτελέσει δηλαδή ένα στήριγμα για τα εθνικά ταμεία καθάρισης. Κάτι ακόμα που θεωρώ πως είναι κάπως περίεργο στην οδηγία δεν υπάρχουν πολλοί περιορισμοί όσον αφορά τις δυνατότητες κάθε χώρας να οργανώσει το Ταμείο Εκαθαρίσεων ή εξαγοράς τραπεζών Ε, και ενώ δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο ε, μεσοπρόθεσμο ταμείο που να καλύψει αυτές τις ε, περιπτώσεις. Επίσης, αν περάσουμε στο σώμα των εποπτών και στην περίπτωση της Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σχέση αυτή που συμπεριλαμβάνει την έγκαιρη, την πρώιμη μάλλον παρέμβαση αλλά και τεράστιες δυνατότητες παρέμβασης, πώς αυτό συνδυάζεται με τη μεταφορά των υποθέσεων σε εθνικές, εθνικά σώματα ε, καθάρισης πώς θα συνδέσουμε τις δύο φάσεις ώστε να μην αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου οι εθνικές αρχές έχουν λόγο ενώ μετά την παρέμβαση ε, την ενδεχόμενη του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην προχωρήσουν μέχρι τέλους όσον αφορά τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Πώς θα υπάρξει δηλαδή στενότερη σύνδεση ανάμεσα στις δύο ε, φάσεις. Το Κοινοβούλιο θέλει να ξεχωρίσει τα προγράμματα εγγύησης των ε, καταθέσεων από το, τα ταμεία εκαθάρισης. Ε, εμείς έχουμε την ε, αντίληψη ότι τα ταμεία εγγύησης καταθέσεων θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία του Βερολίνου, γιατί αν, την, του, του με συγχωρείτε, γιατί στην ουσία θα πρέπει να πληρώσουν δύο φορές. Δηλαδή θα πληρώσουν και για την φάση καθάρισης, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούν και τις καταθέσεις. Όταν θα δούμε πώς θα κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία, ίσως θα μπορούσαν να διοργανωθούν διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως για την ώρα δεν μπορώ να δω ξεκάθαρα ποια είναι η πρόταση για την κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Μάριο, θες να απαντήσεις. Ναι, να απαντήσω σε ένα δυο. Άκουσα τι λέει το Κοινοβούλιο και η γραμμή του Κοινοβουλίου είναι ο διαχωρισμός των, των Ταμείων Εγγυήσεων από τα Ταμεία Εκαθαρίσεων. Εγώ αναφέρθηκα στην μη διάκριση στην μη διαχωρισμό της συζήτηση ανάμεσα στα δύο, γιατί αν, ακόμα και αν τελικά καταλήξουμε σε δύο διαφορετικά ταμεία και σίγουρα υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ αυτού και μάλιστα και στη δική μας αρχική πρόταση υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην ε, χρειάζεται ας πούμε τα ταμεία να πληρώνουν αδίκως ή δύο φορές. Ακόμα και αν λοιπόν καταλήξουμε σε δύο διαφορετικά χωριστά ταμεία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε και τη συζήτηση από αυτού, γιατί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο είναι μεγάλη. Για το, θέμα, το ερώτημα για τους περιορισμούς για τα διάφορα εθνικά ταμεία καθάρισης ή εξαγοράς. Πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες ώστε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς και ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σπάσουμε το δεσμό ανάμεσα στο κρατικό χρέος και, την, και τις τράπεζες. Εδώ ρωτήσατε αν έχουμε διαφωνίες. Ίσως να διέκρινα μια διαφορά με τον καθηγητή Φράνκε. Δηλαδή το θέμα της επικουρικότητας και του κατά πόσο θα πρέπει απολύτως να αποκλείονται κάποια, κάποιοι στόχοι επειδή δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας. Ε, λέω ίσως να έχουμε διαφορά γιατί το, ανείχνευσα μια ενδεχόμενη διαφορά, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα με καλούς εναρμονισμένους κανόνες και επιπλέον κάτι ακόμα ίσως. πάντως ο αποκλεισμός ε, του πεδίου για τη μια ή την άλλη τράπεζα θα είναι πάντα δύσκολη. Ο Ντάνιελ θέλει να παρέμβει. Υπάρχει πάντα διαφορά τεχνικά μεταξύ τράπεζας και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Υπάρχουν παραδείγματα κάποιων ομίλων, η Rai, η και η Drabobank στις κατοχώρες. Υπάρχουν πολλές θυγατρικές τράπεζες, αλλά οι απόπτες αντιμετωπίζουν ως ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, διότι στην πραγματικότητα ο ένας εγγυάται για τον άλλον. Και η λύση για τις τράπεζες στη Γερμανία είναι για τον ε, σκοπό της εξυγίασης να θεωρούνται ως ένα. Να υπάρχει λοιπόν ένας ε, κίνδυνο, γιατί ο καθένας εγγυάται για τον άλλον. Να υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνο δηλαδή και νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσαμε να το χειριστούμε έτσι. Όχι εύκολα, αλλά τουλάχιστον ενοιολογικά ε, ως σύνολο. Όσον αφορά τώρα... για την εποπτεία. Σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, δεν ξέρω τι γίνεται ε, σε καθημερινό επίπεδο. Ε, πώς αποφασίζονται το κλείσιμο μιας τράπεζας, το κλείσιμο των λογαριασμών, ε, τι γίνεται από εκεί και πέρα όταν τα εθνικά κονδύλια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά λοιπόν τα οποία δεν έχουν νόημα από αρκετά πρίσματα αν εξετάσουμε την ταμιευτήρια στην ε, Γερμανία για παράδειγμα και τα εξετάσουμε ως σύνολο θα πούμε ότι η ευθύνη για τις τράπεζες έχει ανέβει προς τα πάνω και επομένως όταν κάτι πάει στραβά η ευθύνη θα πρέπει να είναι άνωθεν δηλαδή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης. Ε, ε ακόμα και αν έχετε ένα ταμείο εξυγίανσης ή όπως αλλιώς θέλετε να το αποκαλύψετε. Ε, σκεφτείτε το σύστημα, όπως είπε και ο ε, ε, Μάριο. Εάν περάσει αυτή η έκθεση Λικάνεν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε το σύστημα DGS για την εγγύηση των καταθέσεων μέσω του Ταμείου Εξυγίανση και θα έχουμε και κάτι ακόμα για το υπόλοιπο τμήμα των τραπεζών. Σε γενικέ γραμμέ όμω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, το παράδειγμα του FTIC στι Ηνωμένε Πολιτείε που κατάφερε επιτυχώ να αντιμετωπίσει αρκετέ περιπτώσει ε, όπου είχαμε κινδύνους ε, ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν του κινδύνους σε συστημικό επίπεδο στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά μπόρεσαν να επιλύσουν κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ε, στην Ιρλανδία βέβαια δεν είχαμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Και τέλος, για το, ε, το ESM δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα είναι εκεί για να μπορέσουμε να λύσουμε κάτι άλλο. Δεν θα δεχόμαστε τα ομόλογα και τα υπόλοιπα των τραπεζών δεν θα έχει την ίδια διαδικασία με τις εθνικές τράπεζες. Θα βλέπουμε τι γίνεται όταν τα ε, κλασικά συστήματα της εγγύησης των καταθέσεων και των ε, ταμείων των εξυγίανσης δεν, μπορούν να έχουν, δεν έχουν αρκετά κονδύλια, που είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως. Και άλλα μέλη θέλουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τους δώσω το λόγο. Ξέρω ότι ο κύριος Λάγκρεν ήθελε να απαντήσει και σε κάτι. Θα μπορούσαμε ε, να σας δώσουμε το λόγο να απαντήσετε σύντομα, διότι το πάνελ είναι ο Ντάνιελ και ο Μάριο. Σύντομα λοιπόν, αν θέλετε, απαντήστε. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, το FTIC και ε, το σύστημα στη Σουηδία, όπου θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ε, ταμεία καταθέσεων, κονδύλια καταθέσεων ε, να χρηματοδοτούν άλλα προβλήματα παρά να αναλαμβάνεται το κόστος από άλλους φορείς. Θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Νομίζω ότι και άλλοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ανταλίν, Πίτερ, Γκούναρ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Κύριο Σάντσες Πρεσέδο. Εγώ νομίζω ότι οι κίνδυνοι σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με εθνικά δίκτυα. Αλλά οι διασυνοριακοί κίνδυνοι χρειάζονται μηχανισμούς διασυνοριακούς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. και νομίζω ότι αφορά μια συζήτηση που δεν ε, γίνεται μόνο εδώ, γίνεται και στις Ηνωμένε Πολιτείες αν υπάρχουν ε, συστημικοί φορείς ή φορείς που ε, εντάσσονται σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό και κάποιοι μικρότεροι που δεν ε, εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να έχουμε πρόβλημα ίσων όρων ανταγωνισμού. Και το θέμα είναι κατά πόσον θεωρούμε ότι τους διασυνοριακούς κινδύνους θα πρέπει να τους ε, έχουμε με μηχανισμούς ε, εξυγίασης, ε, γιατί να εξετάσουμε μόνο το bail-in και να μην έχουμε και το bail-out. Διότι εάν έχουμε bail-in σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε bail-out σε εθνικό επίπεδο. Äh, ναι, στη τελευταία παρατήρηση να πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά το σχήμα εγγύηση των καταθέσεων, έχουμε θέσει κάποια όρια μεγέθους και πιστεύουμε εδώ ότι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το σχήμα εγγύησης των καταθέσεων έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει διάσωση εδώ χρειαζόμαστε από ό,τι φαίνεται μια επιπλέον λύση για μεγάλες τράπεζες που δεν καλύπτονται με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και παρόλα αυτά χρειάζονται διάσωση. Αυτό είναι νομίζω το θέμα. Πρόκειται για μια ευελιξία ελευθερία σε εθνικό επίπεδο και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το πολύ θεσμοθετημένο σύστημα, εμείς σαν κοινοβούλιο εδώ Έχουμε δώσει δυνατότητες, εργαλεία στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσουν σε εθνικό επίπεδο για μικρές και μικρομεσαίες τράπεζες να βρουν λύσεις. Όσον αφορά τον κίνδυνο των α, ταμιευτηρίων, πως τη πάρκασε; εγώ νομίζω ότι όσον αφορά τους κινδύνους δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνεταιριστικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι τα ταμιευτήρια στη Γερμανία τουλάχιστον έχουν τελείως διαφορετική μορφή από αυτή άλλων κρατών. Υπάρχει περιφερειακός χαρακτήρας, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει μόνιμος έλεγχος και υπάρχουν εγγύησει ότι αυτός ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος, μικρός. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν πολλοί και κατακαιρματισμένοι ε, κίνδυνοι, μικροί, περιορισμένοι, έτσι ώστε το σύστημα αμέσως να εντοπίζει το πρόβλημα και να μπορεί να το ε, αντιμετωπίσει πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γι' αυτό και θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να δούμε με διαφορετικό τρόπο αυτές τις περιπτώσεις. Ο Γκούναρ. Τώρα ή αργότερα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά τον κύριο Γκρός. Πώς καθορίζεται ο συστημικός κίνδυνος από εθνικό επίπεδο, κάτι που είναι συστημικό σε εθνικό επίπεδο είναι για όλη την οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το πρόβλημα των ισπανικών τραπεζών. Ποιε είναι οι επιπτώσει για τι γερμανικέ, τι γαλλικέ ή το ίδιο μπορούμε να πούμε για τι ελληνικέ τράπεζε. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια εθνική αντιμετώπιση, μπορεί να υπάρξει και ένα ευρωπαϊκό ταμείο για την εξυγίανση και τη διάσωση και το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν επικαλύψεις. Ίσως να είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο, αλλά καθολική λύση δεν είναι. Όπως είπε κάποιος από τους ομιλητές, μπορεί να υπάρχουν τελικά συστήματα διάσωσης, αλλά ποιος πληρώνει σε τελική ανάλυση ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Και θα πρέπει να ορίσουμε κανόνες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δημόσια παρέμβαση, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση όπου τελικά κινδυνεύει να πληρώσει ο φορολογούμενος χωρίς αυτό να είναι η ίστατη λύση. Με πολύ συγκεκριμένους κανόνες και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό. Γιατί στην πράξη και τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Να επανέλθω στο Μάριο, στον Ντάνιελ, στον καθηγητή, τον κύριο Φράγκε. Όσον αφορά την εγγύηση των καταθέσεων καταρχήν. Μάριο, ευχαριστώ. Στην ερώτηση του πρώτου μιλητή, τα τελευταία δύο χρόνια εγώ πάντα δύσκολα μπορώ να διακρίνω τι είναι εθνικός ε, κίνδυνος και τι είναι υπερεθνικός κίνδυνος. Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα που φαίνονται να είναι εθνικά, έμεσα ή άμεσα, έμεσα ή άμεσα, επαναλαμβάνω, γιατί έχουν συνέπειες. Παραδείγματο χάρη στο κρατικό χρέος, βλέπουμε ότι ξεπερνούν τον εθνικό κίνδυνο. Πριν από δύο ή τρία χρόνια θα σας είχα πει τι πιστεύω και η άποψή μου θα ήταν πιο εύκολο να βασιστεί σε μια διαχωριστή γραμμή η οποία σήμερα για μένα δεν ισχύει πια. Το θέμα τώρα το ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να υπάρξει η παρέμβαση. Διαπιστώσατε όλοι ότι υπάρχει ευρεία αναγνώριση για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί το επίπεδο και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του μηχανισμού εναρμονισμένων κανόνων. Τώρα, το σύστημα αυτό που προτείνουμε για τον Μπέιλιν είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει για πολλές κατηγορίες τραπεζών. Κάποιοι προτείνουν πολύ λίγα προϊόντα και τράπεζες. Αυτά όμως μπορεί να προσαρμοστούν και σε πολύ μεγάλες τράπεζες και σε μεσές τράπεζες ή και άλλες τράπεζες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει ένα επίπεδο όχι μόνο που καλύπτει πολλές χώρες, αλλά καλύπτει και πάρα πολλές κατηγορίες τραπεζών. Και αυτό θα ήταν η απάντησή μου. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, το μέγεθος εκ των προτέρων είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Καθότι πολλά από αυτά που κάνουμε θεωρώ ότι αν λειτουργήσουν θα μειωθεί η πιθανότητα ανάγκης να προστρέξει κανείς σε αυτό το ταμείο ή στο μέγεθος χρηματοδότησης. Το μέγεθος λοιπόν ενός ταμείου είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Παρ' όλα αυτά σε κάποιες από τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες όπως ε, αυτό που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να μην αρκεί το ποσό που έχει προβλεφθεί και να πρέπει να εφευρεθούν άλλες λύσεις. Ο Ντάνιελ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, να πω κάτι για τα ταμιευτήρια, τα Sparkassen. Υπάρχει διαφορά μεταξύ χαμηλού κινδύνου ως όμιλος ή αν είναι ένας ο κίνδυνος ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι κατ' ουσίαν είναι ένας ο κίνδυνος. Τώρα μεγάλος ή μικρός, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αν η διαχείριση είναι πολύ καλή, μπορεί να είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος. Και τότε βέβαια θα φαίνεται στην αξιολόγηση κινδύνου και στο κόστος χρηματοδότησης και εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά για ένα ταμείο εξυγίανσης θα είναι ένας ο κίνδυνος σίγουρα. Συμφωνώ με τον Μάριο που λέει ότι δεν έχει νόημα να πούμε διαφορά μεταξύ εθνικού και διασυνοριακού κινδύνου. Και όπως λέγαμε υπάρχουν εθνικά προβλήματα που είναι συστημικά στην Ευρωζώνη σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του φαινομένου του ντόμινο. Χωρίς διασυνοριακό υπάρχει ένας ε, εθνικός κίνδυνος, επηρεάζει το κράτος, καταραίει το κράτος και έχουμε το φαινόμενο ντόμινο. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε Ευρωπαϊκό Ταμείο η πιθανότητα δεν είναι ποτέ μηδενική δεν είναι μηδέν, αλλά η πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα σε εθνικό επίπεδο και να δώσει ε, το έναυσμα στο φαινόμενο ντόμινο θα μειωθούν πολύ. Σίγουρα δεν υπάρχει βεβαιότητα στην ζωή, εκτός αν υπάρχει ε, χρηματοοικονομική κρίση αλλού. Αλλά η δυνατότητα ε, αντιμετώπισης των μεσαίων κινδύνων αυξάνεται πολύ, βελτιώνεται. Επίσης θα έλεγα ότι οποιοδήποτε ταμείο εξυγίανσης για όλη την Ευρωζώνη θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανθεκτικό, πολύ πιο στιβαρό. Σε εθνικό επίπεδο λέμε τι θα γίνει αν αφήσουμε αυτή την τράπεζα να καταρρεύσει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είμαστε πιο ε, σκληροί και ανθεκτικοί, να έχουμε γιατί η πολιτική πίεση θα αποδυναμωθεί πολύ όλων αυτών που θα μετέχουν στο bail-in. Ε, δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική διαφοροποίηση. αυτά που κάνει η Κομισιόν, αυτά που μπόρεσε να προτείνει μέχρι τώρα, συγγνώμη Μάριο, δεν θα πετύχουν πολλά πράγματα. Πρέπει να, γιατί την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να τη μεταθέσουμε στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Δηλαδή, λες ότι θέλεις οικονομική διαφοροποίηση, ενώ δεν θες πολιτική γιατί θέσε να παραμείνουν οι πιέσει σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, δεν είναι κάποια... Δεν το αποσυνδέεις λίγο. Βέβαια καταλαβαίνω που το πας. Ο καθηγητής Φράνκε, ο Πίτερ Σίμονς, έφυγε που έκανε την ερώτηση για τα ταμιευτήρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι μας ακούν θα, τα, ε, πάρουν απάντηση. Τώρα, να ξεκαθαρίσω αυτό για το Ταμείο Εξυγίανσης. Πάντα χαίρομαι αν βλέπω ένα μηχανισμό της αγοράς να δουλεύει παράλληλα με τον πολιτικό μηχανισμό. Και ποιος είναι ο μηχανισμός αγοράς στις, στο γερμανικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τον τραπεζικό. Έχουμε, ε, τομέα, ε, έχουμε τρεις τομείς επιμέρους που υπόκειται σε αυστηρά συστήματα παρακολούθησης γιατί κάθε τράπεζα είναι υπεύθυνη για τι συζημίε των άλλων τραπεζών. Έχουμε αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης λοιπόν και αυτό σημαίνει ότι η ιδέα είναι να έχουμε τραπεζικές ενώσει που θα ε, έχουν το δικό τους δίχτυ ασφαλείας, θα το έχουν φτιάξει παράλληλα με την παρακολούθηση μέσα στο δίχτυ ασφαλείας. Οπότε αυτό το δίχτυ ασφαλείας θα δέχεται όσο είναι δυνατόν τις ζημίες και πέραν αυτού του ορίου μπορεί κανείς να σκεφτεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης. Δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε εθνικό Ταμείο εγγύησης, ε, στη μέση, γιατί μετά θα έχουμε αυτή, αυτή τη στενή σχέση μεταξύ κυβερνήσεων και τραπεζών. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όμως τις ενώσεις τραπεζών να επεκτείνουν τα ιδιωτικά τους ε, ταμεία εξυγίανσης και ε, δίχτυα ασφαλείας ο Ντάνιελ. Ερώτηση προς τον ε, παρακαθήμενό σας. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό πανευρωπαϊκά. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να είναι ευρωπαϊκό, μπορεί να είναι και σουηδικό. Δεν, δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι πανευρωπαϊκό. Θες όμως διαφοροποίηση κινδύνου. Θέλω παρακολούθηση σε ιδιωτικό επίπεδο, τι ιδιωτικές τράπεζες, από την Ένωση Τραπεζών, Καλώς. Να δούμε όμως, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, είναι εφικτό. Ξαναγυρίζομαι στα συστημικά αποτελέσματα. Έχουμε παράδειγμα μιας χώρας που έκανε αυτό στην κρίση την τωρινή. Η Δανία ε, πλήγει πολύ νωρίς και σκληρά στον τραπεζικό τομέα και πλήρωσαν όλες οι τράπεζες. Ο τραπεζικός τομέας ε, πλήρωσε για να ε, καθαριστούν οι πιο αδύναμες τράπεζες που ήταν αρκετά σημαντικές. Το κράτο δεν πλήρωσε, οι φερολογουμένοι δεν πλήρωσαν. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι προποτίθεται η ύπαρξη πολύ ισχυρών τραπεζών που θα βοηθήσουν τι αδύναμε. Δεν θα είναι συστημική κρίση αυτή τότε. Δεν ξέρω πώ θα την πείτε. Δεν νομίζω να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, η ιδέα του να ε, βάλουμε το βάρος ε, στις ισχυρές τράπεζες για να διασώσουν τις αδύναμες είναι κάτι που πρέπει να τα αποφύγουμε στο μέλλον. Επίσης στη συζήτηση αυτή πρέπει να θυμόμαστε ότι με όλα τα νομοθετήματα τώρα ο τραπεζικός τομέας ε, θα έχει πραγματικό κεφάλαιο 20 με 25%. Είναι τελείως διαφορετικό το σενάριο αυτό και όλη η ακαδημαϊκή έρευνα υποδηλώνουν ότι θα μειωθεί το κεφάλαιο στο 1 δέκατο αυτό που ήταν πριν από την κρίση. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι χαμηλότερη, η συχνότητα θα είναι μικρότερη και το εύρος των ε, επεισοδίων θα είναι ε, πιο περιορισμένο. Τώρα, για τους επόπτες ε, εθνική έναντι ευρωπαϊκών, ευρωπαίων. Εδώ θα περιπλακούν τα πράγματα. Τοπική εποπτεία, ευρωπαϊκή εποπτεία ε, τα, στα σώματα θα μετέχουν και τοπικοί επόπτες και διασυνοριακοί, αν είναι ε, μια μικρή τράπεζα που να έχει διασυνοριακές συναλλαγές και μπορεί να έχουν επόπτη ο οποίος θα βρίσκεται σε χώρα εξωτερική και θα, θα, έχουν ταυτόχρονα και μια μεγάλη τράπεζα στη χώρα που εδρεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε θα έχουμε ευρωπαϊκά ε, ε, κεφάλαια και τοπικά και θα έχουμε μια Ευρώπη ε, δύο επιπέδων, πράγμα που θα περιπλέξει πάρα πολύ την κατάσταση. Πράγματι. Γκούνταρ, νομίζω ότι επαφίεται σε σένα να κάνεις είτε κάποιες τελευταίες ερωτήσεις είτε να ολοκληρώσεις τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εξαγάγουμε τα, πιο πραγματικά, τα πραγματικά και τα πιο ευφύ συμπεράσματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η συζήτηση και από ό,τι είδα ήταν εύκολο να διαφωνεί στο πάνελ, ειδικά στο τελευταίο τμήμα της συζήτηση και όχι στην αρχή και τόσο. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. ένα ε, τα οποία αναφέρθηκαν ε, στο τέλος αυτής της συζήτησης είναι κατά πόσον αυτή η χρηματοδότηση εξυγίασης θα γίνεται εκ των υστέρων ή εκ των προτέρων. Και είναι πολύ σημαντική η διαφορά μεταξύ εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Παρά το γεγονός ότι αν ε, γίνει εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι έχουμε χρήματα. Ενώ αν γίνει εκ των υστέρων δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Όμως αν γίνει εκ των προτέρων είναι μια μορφή ασφάλιση εκ των υστέρων σημαίνει ότι όσοι συμπεριφέρθηκαν καλά θα πληρώσουν για αυτού που δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά. Και εγώ αυτό πραγματικά το αποκαλώ ηθική επίθεση. Επειδή κάποιο είναι τράπεζα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει ε, για αυτόν που δεν συμπεριφέρεται καλά στην όλη, ε, στον όλο κλάδο, διότι τότε θα πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα στην κοινωνία. Οι καλέ επιχειρήσει θα πρέπει να πληρώνουν για τι κακέ επιχειρήσει και οι καλοί βουλευτέ θα πρέπει να πληρώνουν για του κακού. Και ο καλό διευθυντή τράπεζα ε, για τον κακό διευθυντή τράπεζα και νομίζω ότι αυτό το σκεπτικό είναι λάθο. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην τη στιγμή όταν τα προβλήματα θα έχουν οξυνθεί, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δράσουμε ε, άμεσα. Και αυτό νομίζω είναι αυτό το οποίο υφέρπει από όλα όσα ακούσαμε από όλους όσους μίλησαν σήμερα στα πάνελ. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που θα έχει νομική σαφήνεια, αλλά ταυτόχρονα θα ε, μπορεί να αντιμετωπίσει και... Ε, ε κάθε κατάσταση όπως ε, τη βλέπει και να είναι ανοιχτή και σε ε, αυτοσχεδιασμούς ε, εντό εισαγωγικών. Οτιδήποτε και να κάνουμε θα προκύψει μια χρηματοπιστωτική κρίση όπως είπε κάποιος από τους ομιλητές σήμερα και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την ευελιξία να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία θα χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και νομίζω ότι με αυτό θα μπορούσαμε ίσως να ολοκληρώσουμε ε, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε σχεδόν ακριβώς την ώρα μας. Ευχαριστώ όλους και χαίρομαι που για, μια φορά, ε, που για μια φορά δεν θα χρειαστεί να καθυστερήσω τους, συναδε... τους διερμηνείς. Τους ευχαριστώ και για την διερμηνία, Πρόεδρος.